Buenos días. Καλή σας ημέρα. Αν θέλετε παρακαλώ καθίστε. parece, continuamos. Αν θέλετε, ξεκινάμε τη συνεδρίασή μα μετά τη συνάντηση των συντονιστών. Σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση τη ημερήσιας διάταξης. Σε σχέση με την πρώτη εκδοχή της που είχατε λάβει, έχουμε πλέον δύο τροποποιήσεις. Πρώτον, η ψηφοφορία για το πολιετές πρόγραμμα για τον Μπακαλιάρο, έκθεση Βαλέσα, ε, θα ψηφιστεί στην επόμενη συνεδρίασή μας. Συνεπώς δεν θα το ψηφίσουμε σήμερα. Και μετά το σημείο 9 για το πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυριμπάτη της κυρίας Λόεβιν θα το συζητήσουμε αμέσως μετά την λήξη της ψηφοφορίας. Μετά δηλαδή το σημείο 6. Και μετά, στα διάφορα, σας το λέω ήδη από τώρα, αν θέλετε να μείνετε, ε, η έκθεση Γκάλαχερ για τα τεχνικά μέτρα, ε, ε, τα αποτελέσματα δηλαδή του τριμερούς διαλόγου είναι στα διάφορα και θα μας ενημερώσει ο κ. Γκάλαχερ. Μετά, ε, πολύ συχνά βλέπουμε αλλαγές στην μέση διάταξη και αυτό βέβαια βλάπτει τους πάντες. Συνεπώς σας λέω το εξής. Ε, προσπαθώ να είμαι ευέλικτος αλλά θα περιορίσω όσο γίνεται τις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Θα περιοριστούμε μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν πραγματικά σοβαροί λόγοι. Μόνο τότε θα αλλάζουμε την ημερήσια διάταξη. Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται συνήθεια να, ε, να κάνουμε ε, το ό,τι καπνίσει, να το πω έτσι, λέει ο Πρόεδρος, ε, σε οποιονδήποτε ζητά αλλαγέ στη μέση διάταξη. Όχι, θα περιοριστούμε μόνο στις πολύ απαραίτητες αλλαγές από τη στιγμή που η μερίσια διάταξη δημοσιεύεται. Ε, οι διαλλαγές, συνεχείς αλλαγές μας δημιουργούν προβλήματα λειτουργίας, προβλήματα παρουσίας κλπ. Ε, αν δεν υπάρχουν ε, άλλα σχόλια για την ημερήσια διάταξη, περνάμε στο σημείο 5. Όχι, το 5 έχει αναβληθεί. Το 6. Μια γρήγορη ψηφοφορία διανατάσεως της χειρός, αλλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή Συμφωνία Αλληλευτική Σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη κυβέρνηση τη Δανία και τη τοπική κυβέρνηση τη Γρυλανδία αφετέρου. Δεν υπάρχουν τροπολογίε. Ψηφίζουμε το ψήφισμα ω έχει. Περ, κατά, αποχέ, καμία, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Κρίστεσεν. Συγγνώμη, ξέχασα το σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων ε, δύο συνεδριάσεων, όπω πάντα. Εγκρίνονται. Ανακοινώσει του Πρόεδρου δεν έχουμε καμία ανακοίνωση. Περνάμε στο σημείο 9, που είπαμε θα το δούμε μετά το 6. Πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας του Κυριμπάτη. Πρώτη ανταλλαγή σήμερα για τα θέματα του πρωτοκόλλου. Ο λόγος στην κυρία Λέβιν. Okay. Uh, thank you, Chair, and, uh... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για το ότι επισημάνατε ότι ορισμένες φορές δεν είναι και πάρα πολύ βολικό όταν υπάρχουν αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη. Δεν είμαι προετοιμασμένη λοιπόν να το συζητήσουμε ω πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξης, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνω ό,τι το καλύτερο για να το συζητήσουμε. Ήθελα λοιπόν να εκφράσω τις κύριους προβληματισμούς μας ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία αλίας με τον κύριο Μπάτ. Η πρώτη ανησυχία ε, αφορά στη διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον σεβασμό της συμμετοχής του Κυριμπάτη στην ε, συμφωνία PNA και τις ε, υποχρεώσεις που είχε αναλάβει το Κυριμπάτη σε σχέση με την ε, συμφωνία αυτή. Τη συμφωνία που υπογράφηκε το 2010 στην διακήρυξη Κορόρ όπου το Κυριμπάτη προσυπέγραψε μαζί με άλλες οκτώ χώρες του Ειρηνικού για τα θέματα του σχήματος για τα αλλιευτικά, ε, τα σκάφη και τα αλλιεύματα. Να αναφέρω κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής στον ειρηνικό ή να δώσω μια γενική άποψη της κατάστασης στον ειρηνικό. το, νησιωτικό κράτη, κράτος του Κυριμπάτη και ακόμα νησιωτικές χώρες είναι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε ε, όσο και το πλείστον, οι περισσότερε από αυτέ, και κατέφεραν το 1982 να συνέλθουν σε μια συνεργασία του μοναδικού πόρου που διαθέτουν κατά βάση του μόνου φυσικού πόρου που διαθέτουν, που είναι ακριβώς ε, η θάλασσα και η αλία, και είναι τα λεγόμενα προσυπογράφοντα ε, μέλη στην Συμφωνία Νάουρου. Αυτά τα οκτώ μικρά νησιωτικά κράτη έχουν συνολική κατά ε, έκταση 4 ε, εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. 14 εκατομμύρια ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι η τρίτη χώρα της ε, ε παροχής τόνου σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μικρά κράτη τα οποία είναι διασκορπισμένα σε μια τεράστια περιοχή και έχουν τεράστια δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ των ίσων, στο ταξίδι μεταξύ των ίσων αυτών, παρά όμως τις δυσκολίες αυτές κατάφεραν να έχουν ε, μια περιφερειακή προσέγγιση στο μοναδικό μεγάλο περιουσιακό του στοιχεία που είναι ακριβώς τα αλλιεύματα στην περιοχή τους. Ερχόμενοι τώρα συγκεκριμένα στο Κυριμπάτι, έχει 100.000 κατοίκους σε 33 διασκορπισμένα νησιά, εκ των οποίων μόνο τα 21 είναι κατοικημένα. Το ΑΕΠ είναι από τα χαμηλότερα των ε, χωρών, των λιγότερων επιτυγμένων. Ε, κατατάσσεται μία από τις λιγότερο επιτυγμένες χώρες ΑΚΕ βασίζεται πάρα πολύ στις αλλιευτικές, ε, ε άδειες που ε, εκχωρεί σε αλλοδαπές ε, χώρες αλλιευτικές και έχει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την, την Ιαπωνία, Ταϊβάν και την Κορέα και επίσης με κάποιες εταιρείε στον Ισημερινό και το Ελσαλβαδόρο. Και επίσης δέχεται χρήματα από πολυμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μέσω των ΙΠΑ. Οι ΙΠΑ λοιπόν έχουν αλλιευτική συμφωνία πάνω σε περιφερειακή βάση. Κατά βάση δηλαδή δεν διαπραγματεύονται με τα μονομένα τα μικρά νησιωτικά κράτη, αλλά έχουν μια πολυμερή ε, συμφωνία με όλες τις χώρες ε, οι οποίες ε, έχουν τα συγκεκριμένα αυτά αποθέματα τόνων τόνου που προφανώς ταξιδεύουν μεταξύ των διαφόρων αυτών χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγάλος ε, χορηγός ε, της ε, αναπτυξιακή προσπάθειας, αν και δεν περιλαμβάνεται στην σχετική στρατηγική, τη γενική, αλλά παράγεται μέσω του τομεακού τομέα της Συμφωνίας Αλίας, που είναι λίγο παράξενο. 80% των οικοκυριών στο Κυριμπάτι βασίζονται στην Αλία και η χώρα έχει προσδοκίες να ε, εξάγει τόνο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και φιλέτα τόνου. Από το 1996 το Κυριμπάτι μέσω των ΙΠΑ έχει διαπραγματευτεί μια συμφωνία οικονομικής ε, ε, συμφωνίας για να ξεπεράσει τη σχετική προηγούμενη συμφωνία που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Κοτονού που είναι προτιμησιακής σχέσης σύνδεσης. Κατά βάση λοιπόν αυτό που λένε το κύριο είναι ένα εξαιρετικά μικρό και ευάλωτο νησιωτικό κράτος. Έχει πετύχει στην διαπραγμάτευση και τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών με άλλα μικρά νησιωτικά κράτη στα πλαίσια της Συμφωνίας ε, Νουαρού, κράτη του Ειρηνικού δηλαδή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά βάση έχει αρνηθεί να διαπραγματευτεί σε περιφερειακή βάση με τις χώρες αυτές. Αντιθέτως, αν το θυμάστε και ίσως το θυμάται η Επιτροπή αυτή, η Συμφωνία Μικρονησίας είχε ουσιαστικά απορριφθεί από το Κοινοβούλιο. Και γιατί έγινε αυτό. Είναι γιατί ήθελαν να σεβαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προσυπογράφοντα μέλη ε, της Συμφωνίας Ναϊρού και σε ό,τι αφορά το μοντέλο των αλλιευτικών σκαφών και τη συμφωνία σε ό,τι αφορά την αλληλεία ανοιχτή θαλάσσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το ήθελε, επέμενε να έχει διαπραγμα... διαπραγματεύσεις μεμονωμένα με καθένα μικρό από τα μικρά αυτά νησιωτικά κράτη και επέμεινε να βασίσει μια συμφωνία επί τη βάση του, των κόρων και όχι μια συμφωνία με βάση του τύπου των ε, αλλιευτικών σκαφών που η Ρίστον Παρόδο ε, έχει, γίνει, ε, έχει γίνει δεκτό το μοντέλο αυτό από την ε, ε, Παγκόσμια Συμφωνία, στην οποία, ε, τη συμφωνία που έχει γίνει σχετικά με την Αλία από το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και έχει, την οποία έχει προσυπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα λοιπόν, οι ΗΠΑ έχουν αποδεχθεί αυτή την περιφερειακή βάση για τη Συμφωνία της Αλίας, το κ. Μπάτη έχει προσυπογράψει Θα ήθελα να, ξέρω, να ξέρει λοιπόν η, Επιτροπή αυτή ποιες εντάσεις υπάρχουν και τι αντιμαχίες έχουν προκληθεί στην περιοχή. Πριν από λίγους με, ε, μήνες μπορούσαμε να βρούμε σχετικά άρθρα στις εφημερίδες από την περιοχή αυτή όπου ο πρόεδρος της Συμφωνίας Νεαρού ήταν εξαιρετικά επικριτικός για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί το βάρος της, την εξουσία που έχει και την ισχύ που έχει στην περιοχή αυτή για να ουσιαστικά διεμβολήσει και να χωρίσει τους εταίρους της Συμφωνίας Νιαρού. Αντί αντίθετα να επιδείξει την επιθυμία της να διπραγματευτεί σε περιφερειακή βάση, που το κάνει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τις ε, συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας, επιλέγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματεύεται μεμονωμένα με καθένα από τα μικρά αυτά ε, νησιωτικά κράτη του ειρηνικού, που προφανώς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα ε, για τους πόρους, το εισόδημα το οποίο μπορούν να, να ε, ελκύσουν από τις ε, ε, αλλιευτικές συμφωνίες που συνάπτουν με εξωτερικά κράτη, ενδιαφέρονται και για μελλοντικέ συμφωνίες οικονομικής εργασίας και ενδιαφέρονται για την αναπτυξιακή βοήθεια που μπορεί να τους χορηγηθεί. Και ουσιαστικά φαίνεται να υπάρχει μια έλλειψη συνοχής σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή πλευρά, την κοινοτικών πολιτικών και την προαγωγή των περιφερειακών προσεγγίσεων και ουσιαστικά η κοινή αλληλευτική πολιτική αποτελεί αντικείμενο σε περιφερειακή βάση, ενώ οι σχετικές ε, άδειες και πολιτικές περιαλίες γίνονται αλλιευτικής σύμπραξης γίνονται σε μεμονωμένη βάση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αναγνώριση αυτού των, αυτής της συμφωνίας που έχουν επιτύχει αυτά τα μικρά οχτώ νησιωτικά κράτη που προσπαθούν να συνεργαστούν και να έχουν μια πολύ πιο ενιαία και πιο ισχυρή θέση στη διαπραγμάτευσή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση που εξάλλου ουσιαστικά είναι μια, ένας συνασπισμός 22 ε, εξαιρετικά ανεπτυγμένων χωρών και επομένως έχουν πολύ πιο ισχυρές θέσεις στην ε, διαπραγμάτευση από από κάθε έννοια. Η έκθεση αξιολόγησης από τη Συμφωνία Κυριμπάτη καταδεικνύει επίσης αυτή την ε, ασυνέπεια και είναι λίγο παράξενο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο σε σχέση με τις ε, συμφωνίες ε, αφενός αφενός ε, αλληλευτικής ε, συνεργασίας και αφετέρου ε, αναπτυξιακής πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να το γνωρίζει ότι η συζήτηση αυτή είναι εξαιρετικά έντονη αυτή τη στιγμή στον ειρηνικό. Την περασμένη άνοιξη ήμουν μαζί με την κυρία Φράγκα, η οποία μπορεί να τεκμηριώ... η οποία μπορεί να τεκμηριώσει ε, και να υποστήριξω ότι όντω υπάρχει πολύ μεγάλος ε, ε, αντίκτυπος και πολύ μεγάλη αναταραχή στα νησιά εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχεται και, θεωρεί, και θεωρούν ότι έρχεται να σπάσει και να κόψει τους βασικούς τους πόρους και την ενιαία θέση τους που έχουν στην προσπάθεια ελέγχου των πόρων τους. Όπως ξέρετε, η όλη περιοχή εκεί όπου μπορεί κανείς να αλλιεύσει τόνο είναι περίπου ε, ουσιαστικά το 95% της ε, ΑΟΣ των μικρών αυτών ε, νησιών. Άρα πολύ θεμητά και λογικά προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο των πόρων τους. Και το διάχυτο, η διάχυτη αίσθηση εκεί, και ισχύει 100%, η διάχυτη αίσθηση εκεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει ουσιαστικά για να καταστρέψει αυτή τη συνεργασία που έχουν επιτύχει, και χρησιμοποιεί την εξουσία της σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις, την αναπτυξιακή βοήθεια κλπ. για να χωρίσει και να σπάσει αυτό το ενωμένο μέτωπο που έχουν τα νησιωτικά αυτά κράτη. Το ίδιο ισχύει και με τα νησιά του Σολομόντα. Το επισημαίνω λοιπόν αυτό και θα ήθελα να ακούσω σχετικά τις απόψεις των συναδέλφων. Και η ο άλλος μου προβληματισμός, η άλλη μου ανησυχία αφορά την, ε, την βιωσιμότητα των, ε, του εξοπλισμού συγκέντρωσης ε, ηχθείων που πραγματικά θέτησε απειλή τα, τους τα νεογνά και θεωρεί, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος, κάποιος σχετική πρόβλεψη στο πρωτόκολλο συμφωνίας που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής και εκφράζουμε εκπληκτόμαστε ιδιαίτερα που το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει και τα σκάφη με παραγάδια. Ουσιαστικά δεν υπήρχε καθόλου ε, τέτοια πρόβλεψη και τέτοιες σχετικές ε, άδειες στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Φαίνεται λοιπόν τώρα ότι δεν υπάρχει συνέπεια με τους οικονομικούς ε, περιορισμούς ε, του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί δεν είμαι καθόλου πεπισμένη ότι θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον και στο μέλλον, αλλά με πάση περιπτώσει μας, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, διευκρινίσει το ζήτημα και υπάρχουν διαφορετική θέση. Αυτή είναι η κύριοι προβληματισμού μου, στους οποίους ε, διαφωνώ και ευχαριστώ και περιμένω να ακούσω τις απόψεις Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, έχει ζητήσει το λόγο κυρία Φράγα. να ξεκινήσω ε, όπως και η κυρία Λέβιν λέγοντας ότι στην πρώτη έκθεση για, την οποία, για το Κυριμπάτι για την οποία εγώ ήμουν συγγήτρια επί τη ευκαιρία της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειρηνικού είχαμε μιλήσει για την ανάγκη να συγκεντρωθούμε, ε, συγκεντρώσουμε τη δράση μας σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό δεν έγινε όχι για λόγους αλίας τόσο πολύ, όσο γιατί οι τρεις γενικές διευθύνσεις της ε, Κομισιόν, οι ε, θαλάσσιων υποθέσεων ε, και οι άλλες δύο, εμπορίου, trade κλπ, δεν συντονίστηκαν αρκετά. Γιατί οι άλλες γενικές διευθύνσεις εκτός της ΜΑΡΕ δεν καταλαβαίνουν πολύ από θέματα αλίας. Τούτου λεχθέντος και χάρη της αλήθειας, τα πράγματα αλλάζουν και ελπίζω να μας το επιβεβαιώσει η Κομισιόν. Η ίδια η Κομισιόν αντελήφθη ότι ε, με τον τρόπο που ακολουθούσαμε όμως τώρα καταλήγουμε σε αντιφατικές πολιτικές ε, με αυτή την αποσπασματική προσέγγιση που ακολουθούσαμε ως τώρα. Η Κομισιόν λοιπόν αλλάζει την προσέγγιση της και μια και θα είμαι η συγκήτρια για την στρατηγική για τον ειρηνικό, θα ήθελα, λέω, ε, στην Αλία να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση πιο περιφερειακή όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ε, συμφωνία με το Forum Fisheries Agency, το FFA, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από τις διμερείς συμφωνίες. Τούτου λεχθέντος, Η ζώνη αυτή, η περιοχή αυτή είναι η πιο πλούσια ζώνη του κόσμου σε, αποδημητικά, ε, σε αποδημητικούς ηχθείες. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτές οι χώρες ε, είναι θεματοφύλακες όμως αυτής της ζώνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τέσσερα πλοία εκεί. Τέσσερα λευτικά σκάφη. Συνεπώ δεν δημιουργήσαμε εμεί το πρόβλημα στην ε, Περιφερειακή Οργάνωση, μάλιστα αλλία για αυτά τα ύδατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που πιο πολύ υποστηρίζει κριτήρια διαφάνεια. Και ζητά να υιοθετηθούν τα όποια μέτρα χρειάζονται για την καταπολέμηση της άναρχης αλίας, της IUU. Αυτές οι χώρες τι θα έπρεπε να κάνουν σε περιφερειακό επίπεδο. Θα έπρεπε να διαπραγματευτούν, μάλλον εμείς θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε με όλες αυτές τις χώρες μια κοινή συμφωνία, αλλά θα έπρεπε να τους ζητήσουμε διαφάνεια που αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Γιατί η περίφημη συμφωνία Ναούρου, για την οποία αναφέρθηκε η κυρία Λόβιν, επιβάλλει ένα σύστημα που ονομάζεται Vessel Day Scheme. <laughs> Τι σημαίνει αυτό. Σου πουλάω μέρες αλίας χωρίς καμία διαφάνεια γιατί δεν ξέρω πόσες είναι οι συνολικέ μέρες αλεία και ούτε πώς κατανέμονται, έτσι. Σου πουλάω λοιπόν μέρες αλεία. Για κάθε μέρα, κάθε μέρα χρεώνεται 6.000 ευρώ, αλλά δεν υπάρχει κανένα είδου έλεγχος. Με αυτόν τον τρόπο ε, χειροτερεύει η κατάσταση των αλλιευμάτων και των αποθεμάτων κάθε μέρα και δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνία λίγας λοιπόν με, τον, με το που είναι η, συμφωνία, η λύση την οποία έχουμε βρει προς το παρόν έτσι ώστε να συνεχίσουν να αλληλεύουν τα τέσσερα σκάφη μας είναι το μη χείρον βέλτιστον. Η έκθεση αξιολογήση λέει ότι η σχέση κόστου κόστος-οφέλους είναι καλή, πράγματι. Εν γέννη αυτά που αναφέρει η συμφωνία είναι καλά. Ε, Τώρα, σε ό,τι αφορά το κόστος, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση που αυξήθηκε ελάχιστα, ε, το κόστος αυξήθηκε για τους πλειοκτήτε. Και θα σας δώσω ένα στοιχείο γιατί είναι συγκρίσιμο. Παλιότερα ε, πληρώναν οι πλειοκτήτε 21.000 ευρώ για ένα σκάφος ε, με κυκλικά δίχτυα. Τώρα πληρώνει 131.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, η συμφωνία αυτή θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη οικονομικά αποδοτική για το Κυριμπάτι. Και όπω έλεγε η κυρία Λεωβίν, ε, θα έπρεπε οι προσεγγίσει περιφερειακού τύπου όπω αυτέ που, ακολουθούν οι ΗΠΑ θα ήταν καλέ και ωφέλιμε όχι μόνο για τι ίδιε αυτές τις χώρες αλλά και για μα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είναι ωφέλιμε ήδη για τι Ηνωμένε Πολιτείε και για άλλες χώρες που έχουν περιφερειακές συμφωνίες. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στρατηγική θα ακολουθήσει και η Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, η συμφωνία με το Κυριμπάτι είναι ωφέλιμη, αποδοτική και για τα τέσσερα σκάφη μας που βρίσκονται εκεί, αλλά και για το Κυριμπάτι. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρεσέδο. Ο κύριος Πρεσέδο. Συμφωνώ με τα σχόλια που ακούσαμε για το μέλλον. Είναι χρήσιμο να καταλήξουμε σε μια περιφερειακή συμφωνία. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Οπότε δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα κένο στην αλληλευτική συμφωνία. Οπότε η συμφωνία με το Κυριμπάτη δεν είναι ένα καπρίτσιο. Είναι μία από τις πιο παλιές συμφωνίες με τις ε, χώρες περιοχής αυτής από το 2003. Είναι σημαντική η συμφωνία αυτή για τη σχέση μας με το Κυριμπάτι. Οι διευθετής αυτής της συμφωνίας περιλαμβάνουν ένα σημαντικό οικονομικό σκέλος, αλλά η συμφωνία αυτή ε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της γενικότερης ανάπτυξης των σχέσεων με το Κυριμπάτι. Οι αλληλευτικέ λοιπόν σχέσεις εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο σχέσεων με το Κυριμπάτι. Από το 2003 μέχρι σήμερα ε, έχουν υπογραφεί τρει συμφωνίες. Αυτή είναι μια συμφωνία ε, που προβλέπει σημαντική αύξηση του, της οικονομικής αντιστάθμισης. Περνάμε ε, από 425.000 ευρώ στο 1.225.000 ευρώ, σημαντική αύξηση. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τις αλληλευτικές δυνατότητες, να μην δημιουργήσουμε ένα νομικό κενό ε, στις ε, σχέσεις μας με αυτή τη χώρα, υπό την προπόθεση όμως ότι θα καταλήξουμε τελικά σε μια περιφερειακή συμφωνία. Προ τα εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Λέβιν. Η Κομισιόν. Oui, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Λεβίν για την ε, έκθεσή της. Παρουσιάζει πάρα πολύ καλά τα χαρακτηριστικά και τα διακυβεύματα της συμφωνίας αυτής και εν γέννη του ειρηνικού. Καταρχάς, το ζήτημα το κατά πόσο θα μπορούσαμε να πραγματευτεί μια συμφωνία επί περιφερειακής βάσης. Αυτό φανταζόμαστε στην αρχή. Εάν ε, ήταν εύκολο κάτι τέτοιο, και εάν ήταν εφικτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστω θα είχε διαπραγματευτεί επί αυτή τη βάση. Τα πράγματα όμω είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Γνωρίζετε ότι με τα θέματα τη κυριαρχία, ακόμα και αν πρόκειται για μικρά νησιωτικά κράτη, παρόλα αυτά είναι κυρίαρχα κράτη και θίγονται και ζητήματα οικονομικά. Και όταν θίγονται οικονομικά ζητήματα, κάποιο, κάθε κράτος, ανεξαρτήτως μεγέθους, υπεραμείνεται των, ε, των συμφερόντων του. Ε, ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμη μια περιφερειακή συμφωνία, αλλά κατά φαινόμενα καταλήξαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, με τον κύριο Μπάτη, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Αλληλευτικό ε, Στόλο, καταλήξαμε ακριβώς σε αυτή την ε, διμερή συμφωνία. Είπα ότι κατά αυτόν τον τρόπο, με την, συμφωνία, με την συμφωνία με τον κύριο Μπάτη, που δεν ε, εμπίπτει σε μια περιφερειακή βάση και δεν ε, σέβεται όλες τις διατάξεις συμφωνίας ΝΑΓΟΥ. Κατά κάποιο ε. τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ε, διασπάσει το συνασπισμό των κρατών αυτών. Εξαρτάται από την οπτική γωνία που το βλέπει κανείς. Σίγουρα υπάρχει μια ισορροπία, θέλετε, δυνάμεων. Ε, και ένα παιχνίδι συμφερόντος στον ειρηνικό που μπορεί να είναι υπέρ ή κατά κάποιων ε, κρατών. Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως μπορεί να θεωρηθεί μια ενοχλητική ε, ισχύ, μια ισχύ στην ενοχλητική εξουσία γιατί φέρνει μια διαφορετική φωνή στην περιοχή αυτή. Αλλά ανεξαρτήτως των ποιών είναι των διεθνών οργανισμών που είναι στα πλαίσια και στα πλαίσια διμερών συμφωνών, συμφωνιών είτε στα πλαίσια αλληλευτικής πολιτικής στα πλαίσια του ΠΟΕ, πάντα θέλαμε μια ε, συμφωνία η οποία θα ήταν ε, βιώσιμη και, ε, και συμφέρουσα επαμοιβαίω. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά την ε, συμφωνία. Το σύστημα αυτό, ένα σύστημα το οποίο δεν είναι φόρο. Το σύστημα αυτό δηλαδή το οποίο αφορά τα πλαίσια της συμφωνίας αλλιευτικής σύμπραξης που δεν έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και ένα σύστημα το οποίο δεν είναι συνεπές σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των ημερών αλίας. Νομίζω παρόλα αυτά βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας υπεύθυνο εταίρος στην ε, περιφέρεια, ακόμα και αν δεν έχει, ακόμα και αν δεν έχει μέχρι στιγμής ε, υπογράψει συμφωνία παρά μόνο με τον κύριο Μπάτη, ήταν και υπεύθυνη γιατί ε, είναι πολύ σημαντικός αρρωγός της αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγείται στη χώρα αυτή και στις άλλες χώρες της περιοχής. Και όπως η κυρία Φράγκα υπενθύμησε, στην όλη περιοχή δεν έχουμε παρά τέσσερα ε, μεγάλα αλλιευτικά σκάφη. Ε, για Άρα δεν συγκρίνεται αυτό με την παρουσία άλλων αλλιευτικών στόλων, των ΙΠΑ για παράδειγμα ή της Ταϊβάν. Και ως εκ τούτου ο αντίκτυπό μας σε ό,τι αφορά τους ε, υδάτινους ε, υδρόβιους σπόρους είναι πολύ πιο, πολύ πιο Τώρα και σε ό,τι αφορά τα δουλευτικού στόλους έγινε αποδεκτό την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλλεται ένα συγκεκριμένο τίμημα σε σχέση με τα αλληλευτικά σκάφη. Έχουμε αυξήσει τις μέρες αναφοράς για να είμαστε συνεπείς με τα αλλιεύματα και τον τόνο των αλλιευμάτων που παρουσιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και οι εφοπλιστές καταβάλουν πολύ σημαντική ε, προσπάθεια για την έκτακτη φορά και περισσότερα τις ωφέλη που, κατα... που ε, καταβάλουν. Τέλος, ένα τελευταίο σημείο σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για, που αφορούν στη συγκέντρωση αλλιευμάτων, θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακή βάση και σε ό,τι αφορά την, ε, πόσο συνάδει με τη συμφωνία με το Κυριμπάτη, υπενθυμίζω κατά κύριο λόγο ότι είναι ε, ουσιαστικά αναφέρεται στο περισσότερο και είναι σε βάση των, ε, του βάρους των αλλιευμάτων που είναι μόνο το 2% των συνολικών αλλιευμάτων από το στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν έχει τόσο μεγάλη επίπτωση στη συμφωνία την οποία συζητάμε σήμερα, δηλαδή για το νέο πρωτόκολλο ε, για τη συμφωνία αλλιείας που, που συνάπτω μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Μπάτη. So, uh, Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για τις παρεμβάσεις σας. Χαίρομαι που υπάρχει πολιτική συνένεση στο ότι θα πρέπει να έχουμε μια περιφερειακή προσέγγιση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υποστήριξή σας. Είναι πολύ σημαντική. Έχω ακόμα ορισμένα ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πιστεύω πως είναι κάπως παράξενο να λέμε ότι το Κυριμπάτι θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά του και θα επιθυμούσατε να υπάρχει περιφερειακή προσέγγιση. Δεν υπήρχε στην περίπτωση της ε, συμφωνίας για τη Μικρονησία και μάλιστα ήταν καταστροφικό το τέλος διότι οι Μικρονήσοι ήθελαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί την Περιφερειακή Συμφωνία όπως το 2010. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω τι γίνεται με την Συμφωνία για τα νησιά Σολομόντα και ποια είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ίδια? Διότι πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Διότι το Κυριμπάτη είναι η πιο φτωχή χώρα της περιοχής και έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και ήδη εφαρμόζουμε το διέρη και βασίλευε εκεί. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Και νομίζω πως προσπαθούμε να μειώσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένα απειλούμενα είδη. Το 2% δεν είναι πολύ, αλλά το 50% των αλλιευμάτων αφορά είδη που εκεί. Και όσον αφορά τις, ε, τους εξοπλισμούς συγκέντρωσης, δεν έχουμε κάποιο σχέδιο για αυτούς. Ορισμένες φορές αναφερόμαστε στο WCPFC και άλλες φορές δεν το υπολογίζουμε καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τελικά η προσέγγιση μας. Ανέφερα ότι περίπου 50 έως 84.000 ε, είδη καρχαρία είναι παραλιεύματα και ο κυτρινόπτερος τόνος υπεραλιεύεται ή τουλάχιστον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υπεραλίευσης. Επίσης και άλλα είδη τόνου υπεραλιεύονται και υπάρχει μεγάλη, μεγάλος αριθμός ε, ηχθιδίων που παραλιεύονται. Δεν υπάρχουν όρια στον αριθμό του εξοπλισμού συγκέντρωσης που αυτά τα πλοία πρέπει να έχουν. Και η έλλειψη αυτών των ορίων έχει μεγάλες και σοβαρές επιπτώσεις στις συγκεντρώσεις των νυχθείων. Τέλος πάντων όμως, θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να ακούσω τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα νησιά Σολομόντα και για το πώς θα προχωρήσουμε, αποφεύγοντας το Διέρη και Βασίλειο στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λόβεν. Κάτι άλλο, άλλα σημεία. Η Επιτροπή. Η δαγιατή προσέγγιση, αυτή η περιφερειακή, θα ήταν η περιφερειακή, αλλά πάρα πολύ απέχουμε από αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και να διευθετηθούν σε περιφερειακό επίπεδο. Και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πάνω σε αυτό. Και συμπεριλαμβάνεται και το θέμα των ε, συμφωνιών ελιευτικής ε, σύμπραξης. Απουσία όμως συνένεσης και προόδου σε αυτή την περιφερειακή βάση, προφανώς η συνομιλίες κατέληξαν με κάποιες χώρες, όπως έγινε με τη Μικρονησία, με τα νησιά του Σολομόντα, όπου τα νησιά του Σολομόντα θέλησαν να κρατήσουν την αναφορά στο VDS, δηλαδή τις ε, μέρες αλίας, πράγμα το οποίο δεν επιθυμούσαμε και εξήγησα γιατί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η προσέγγιση του να υπάρχει μια συμφωνία αλίας δεν προβλέπεται ε, βραχυπρόθεσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των αλλιευμάτων, θέλω να υπενθυμίσω κάτι, ότι πάνω από το 80% των αλλιευμάτων μας αφορούν d'après l'ensemble des recommandations des scientifiques, une espèce non exploitée, euh, qui n'est pas surexploitée. Ε, αλληλευτικό είδος το οποίο δεν ε, έχει τύχει υπεραλίευσης. Κυρία Φράγκα. Ναι. Θα ήθελα να κοιτάξουν τι κάνουν οι ΙΠΑ ε, και άλλα χώρε σε ό,τι αφορά τη ΣΑΣ, τη Συμφωνία Αλιστικής Σύμπραξης, που έχουν πολύ περισσότερες. Θέλω να θυμίσω ότι είχε γίνει ότι οι χώρες αυτές για τι οποίε μιλάμε απέρριψαν τα, τα προγράμματα διαχείρισης των ε, ΣΑΣ και οι χώρες αυτές ήταν που, που απέρριψαν το σχέδιο διαχείρισης των ΣΑΣ. Καταλαβαίνω λοιπόν την ανησυχία των ε, συναδέλφων, γιατί, αλλά από την άλλη πλευρά ήταν οι ίδιες χώρες οι οποίες απέρριψαν αυτό το σχέδιο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν για το τι λέμε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί όντως να είναι διαλυτική. Είναι όμως από τα λίγα μέλη αυτού του οργανισμού. Γιατί μέλη της ε, οργάνωσης αυτής, όλα τα τι χώρες που αναφέρατε προηγουμένω, δεν έχουν διαφάνεια. Εμείς είμαστε οι μόνοι που υπεραμεινόμεθα κάποιων αρχών, συμπεριλαμβανομένους σε αυτής και του κ. Ζόβεν. Αλλά όπως είπα, ακριβώς αυτές οι χώρες ήταν οι πρώτες οι οποίες απέρριψαν ένα τέτοιο σχέδιο διαχείρισης των ΣΑΣ Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λέβιν, για να τελειώσουμε τη συζήτηση έχει το λόγο. Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρη όμως εάν το Κυριμπάτι αρνήθηκε να έχει σχέδιο διαχείρισης σας στην συμφωνία. Δηλαδή, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ελέγχει τα σκάφη και τη χωρητικότητα, τότε θα έπρεπε να συμπεριλάβει ένα σας στο πρωτόκολλο της συμφωνίας. Δηλαδή, εάν δηλαδή θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι, γιατί να μην υπάρχουν αυτά μέσα στο πρωτόκολλο. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε σε περιφερειακό επίπεδο, μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στο πρωτόκολλο. Ευχαριστώ. Ναι, ε, Νομίζω ότι ε, το συζητήσαμε επαρκώς. Περνάμε στην, στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το 7. Δημιουργία κοινωτικού συστήματο πρόληψη, αποτροπή και εξάλληψη τη παράνομη λαθρέα και άναρχη αλληλεία. Θα θυμάστε ότι στι 6 Σεπτεμβρίου η Κομισιόν υπέβαλε την πρότασή τη. Σήμερα θα κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα. Ο λόγος στον κύριο Ρωμέβα Ιρουέδα. Θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί έχω το κείμενο στα αγγλικά. Ε, είναι θέμα προσαρμογής στην συνθήκη Λισαβόνας, οπότε ε, κοιτάμε ε, τις ε, αρμοδιότητες της Κομισιόν και τις αναθεωρούμε. προτείνονται κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά τον τύπο των πράξεων ε, οι οποίες χρησιμοποιούνται, χωρίς όμως να αλλάζουν οι αρμοδιότητες της ε, Κομισιόν ήρθαμε και σε επαφή με την νομική υπηρεσία που πιστεύει το ίδιο. Συνεπώς γενικά συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες μπορούμε να πούμε ότι η Κομισιόν ε, προτείνει την, ε, ε, την... να υιοθετεί ε, προκράσεις κατεξιοδότηση για θέματα ε, αλλαγής περιόδων πληροφόρηση ε, για θέματα επιθεώρησης φορτώσεων και εκφορτώσεων, επιθεωρήσεων ε, σκαφών τρίτων χωρών. Ε, η για την αποδοχή και την έκδοση πιστοποιητικών ελιευμάτων, για την προσαρμογή της ε, προθεσμίας ε, ανακοίνωσης ε, για την έκδοση των πιστοποιητικών αλλιευμάτων και για την έκδοση ή αναστολή των πιστοποιητικών εγκεκριμένων φορέων εκμετάλλευσης. Σε ό,τι αφορά τις εφαρμοστικές πράξεις, και εδώ έχουμε κάποια θέματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν κάποια ζητήματα. Δεν έχω σαφή ιδέα όμως, γι' αυτό θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Πρώτον, σύμφωνα με τον κανονισμό Γιού, υπάρχει μια πρόταση για μια, ένα κατάλογο των μη συνεργαζόμενων χωρών. Ορισμένα κράτη-μέλη εκφράζουν κάποιου δισταγμού. γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε, ποιες, ποιοι είναι αυτοί οι δισταγμοί και τι μπορούμε να περιμένουμε στη συζήτηση που θα γίνει στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Και ένα δεύτερο ερώτημα, και πάλι είναι ερώτημα, έτσι, έχει σχέση με ένα άλλο κατάλογο, τον κατάλογο των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποτίθεται ότι θα συντάξει και θα διατηρεί η Κομισιόν. Και τα δύο αυτά θέματα εμπίπτουν στο πεδίο των ε, εφαρμοστικών πράξεων. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί, κάποιες απορίες, θα ήθελα να μου πείτε αν έχουμε κάποιες καινούριες πληροφορίες τις οποίες θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Αν βέβαια υπάρξουν σχόλια θα τα λάβω υπόψη μου. Φράγα. Κυρία Φράγα, δύο πραγματάκια. Καταρχήν, διαβάζοντας ε, την ε, πρόταση, έχω κάποιες αμφιβολίες. Πρώτον, για τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται με, κατεξιο... με, πράξη όπως πάντοτε. Νομίζω ότι αυτό υποστεύει και η νομική υπηρεσία. Δεύτερον, για την έκδοση πιστοποιητικών. Για παράδειγμα στο άρθρο 6. Το ανέφερα και σε σχέση με μια ερώτηση που θέλω να υποβάλω στην Κομισιόν. Το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους ε, υιοθετήθηκε η συμπερίληψη νέων χωρών στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων χωρών. Καμπότζη, Φίτζι, Μπελίζε, Παναμά, Σριλάνκα, Τόγκο, και Βανουάτο. Στην ε, ε, συνάντηση της 23 Οκτωβρίου, 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες με τα κράτη-μέλη, όταν διαβάστηκε αυτός ο κατάλογος, το Ηνωμένο Βασίλειο διαφώνησε για τον Μπελίζε, κάτι που με εκπλήσει κύριε Στίβενσον, Ορισμένα κράτη-μέλη είπαν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 18. Αν δηλαδή δεν είναι συνεργάσιμα, θα πρέπει να απαγορευτούν οι εισαγωγές από αυτά τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν ε, και πάλι υπαναχώρησε και είπε δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο κλπ. Οπότε θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα, πού βρισκόμαστε, σε ποια φάση βρισκόμαστε. Γιατί κάθε φορά που ε, βλέπουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ε, αυστηρά ο κανονισμός 1005, η Κομισιόν υπαναχωρεί και δεν εφαρμόζεται, δεν συμμορφώνεται με τον ίδιο τον κανονισμό της. Εφόσον είναι... Βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά έχει σχέση με τον κανονισμό 1005. Τι θα κάνει η Κομισιόν με αυτέ τι χώρε, οι οποίε θεωρούνται μη συνεργάσιμε χώρε. Και γιατί η Κομισιόν αποφάσισε να μην εφαρμοστεί το άρθρο 18. Νομίζω είναι το εδάφιο 1 του άρθρου 18, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υποχρέωση ε, απαγόρευση εισαγωγών από αυτέ τι χώρε. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Μία ακόμα φορά βλέπω η Κομισιόν να μην εφαρμόζει τον ίδιο τον κανονισμό. Ευχαριστούμε κυρία Φράγα. Κανεί άλλο δεν ζητά το λόγο. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. για τα δύο αυτά θέματα. Καταρχάς, για την κατάσταση με τις μη συνεργαζόμενες χώρες και με, με τον κατάλογο των σκαφών παρανομής λαθρέας και άναρχης Όσον αφορά τις χώρες, αυτές τις 8 χώρες που ανέφερε ο συνάδελφος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία μιας πρότασης. Βασικές αρχές που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η διαδικασία γίνεται σε στάδια και αυτό είναι το πρώτο στάδιο και σύμφωνα με τους βασικούς ε, κανόνες του κανονισμού το πρώτο στάδιο με τις τρίτες χώρες είναι να ειδοποιηθούν καταρχάς οι χώρες αυτές για την πιθανότητα να θεωρηθούν μη συνεργαζόμενες. Να λάβουν όλα τα στοιχεία, όλες τις σχετικές πληροφορίες και να προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί ένας διάλογος για επίλυση του προβλήματος. Μέσα στο Νοέμβριο, σε αυτό το μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να υιοθετήσει μια τέτοια απόφαση και το Κοινοβούλιο θα λάβει λεπτομερές σημείωμα που θα αναφέρεται σε όλες τις λεπτομέρειες και στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Το άρθρο 18.1g αναφέρεται στην άρνηση πιστοποίησης αλλιεύματος για τις μη συνεργαζόμενες χώρες βασίζεται στον κανονισμό για την ε, παράνομη λαθρεία και αναρχία αλλά δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτό το έγγραφο μας, διότι το άρθρο 81G ζητά μία απόφαση για πιστοποίηση της χώρας ως μη συνεργαζόμενη. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο ακόμα. Το άρθρο λοιπόν 81G δεν μπορεί να εφαρμοστεί. στις αποφάσεις που θα λάβει η Κομισιόν. Τώρα, όσον αφορά τον κατάλογο των σκαφών, η δεύτερη ερώτησή σας, αν δεν κάνω λάθος, Προβλέπεται η πιθανότητα αυτή όπως γνωρίζετε. Νομικά είμαστε πρωτοπόροι παγκοσμίω. Δεν γνωρίζω να υπάρχει άλλη χώρα που να έχει αυτό το σύστημα. Το σύστημα είναι πολύ καινούριο. υπάρχουν διάφορες νομικές διαδικασίες. Η νομική διαδικασία είναι πολύ περίπλοκη και εμείς εργαζόμαστε πάνω σε αυτές και ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα με, την, ε, με τις ε, διαδικασίες έρευνας. και να ασχοληθούμε με το νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μία πρόταση. Όμως αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, θα διαρκέσει αρκετό χρόνο, διότι είναι περίπλοκη, νομικά περίπλοκη και επίσης διότι είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα ξανά. Σε εκείνη τη συνάντηση σύμφωνα με τις ε, πληροφορίες μου, που μπορούν και αυτές να διαψευστούν βέβαια, ε, νομίζω ότι εγκρίθηκε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αυτές οι 8-9 χώρες στις οποίες αναφέρθηκα. Και δεδομένου ότι αυτό έγινε, αν έγινε, εφαρμόζεται αυτόματα το 18F. Δηλαδή, άπαξ και βρεθούν στην, στον κατάλογο, μπορεί να ζητηθεί αμέσω η, ε, να ζητηθεί αμέσως η απαγόρευση των εισαγών. Τότε όμως διαφώνησαν διάφορες χώρες που βρισκόντουσαν στη συνεδρίαση και τότε η Κομισιόν αντελήφθη ότι ε, δημιουργήθηκε ένα σχετικός χαμός και δεν ήθελε. Αυτό όμως δεν με βρίσκει σύμφωνη, γιατί ε, εφόσον έχουμε εγκρίνει τον κανονισμό, θα έπρεπε να εφαρμοστεί στη διακριμένη περίπτωση το άρθρο 18F. Η Κομισιόν γνωρίζει πολύ καλά ότι χώρε όπω ο Παναμάς, γιατί σε άλλε χώρε δεν είμαι τόσο σίγουρη, αλλά ε, ζητούμε από τον Παναμά μέσω διαπραγματεύσεων να διορθωθεί η κατάσταση. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, ότι η Κομισιόν δεν θέλησε να εφαρμόσει το 18F του 2005. Όμως, οι χώρες αυτές έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον κατάλογο και αφού συμπεριλήφθησαν ετέθη το θέμα της απαγόρευσης και τα κράτη-μέλη διαφώνησαν και τότε η Κομισιόν, όπως είπα, έκανε πίσω. Είναι προφανέ ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση εφαρμογή αυτού του κανονισμού και έχω βαρεθεί πια να μην εφαρμόζεται ποτέ αυτό ο κανονισμό. Δεν θα έπρεπε να απαγορεύσουμε τι αγωγέ σε απορισμένε χώρε για να μάθουν, για να λειτουργήσει ω ε, δίδαγμα και να μάθουν και οι υπόλοιπε. Ευχαριστώ, η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι και η Επίτροπος και η Επιτροπή λαμβάνουν την εφαρμογή του κανονισμού πολύ σοβαρά υπόψη. Και αυτό που κάνουμε στα πλαίσια αυτού του πρώτου καταλόγου των χωρών που θα ειδοποιηθούν είναι, όπως είπα, το πρώτο βήμα. Έτσι προβλέπει η διαδικασία σταδιακά βήματα Και από το 2008, από την αρχή, έγινε ξεκάθαρο ότι ο κανονισμός αυτός που εγκρίθηκε συνδέεται άμεσα με μια μαύρη λίστα και επίσης να πω ότι είμαστε εναρμονισμένοι με αυτά που ήδη έχει δεχτεί το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον έλεγχο για τα αλλιεύματα σκουμπριού. Θα ενημερωθείτε επίσημα με σημείωμα και όπως ε, είπα και πριν, σε αυτό το μήνα θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Θα ήθελε ο εισηγητής να ρωτήσει, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο καιρό θα διαρκέσει, αλλά αν μας διαβεβαιώνετε ότι θα γίνει μέσα σε ένα μήνα, εντάξει. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη, Σημείο 8. Τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο ΣΚΑΙΡΑΚ και τροποποίηση του κανονισμού 850 του 98 και του κανονισμού 1342 του 2008. Θα προβούμε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η συγητής είναι ο κύριος Κούν. Του δίνω το λόγο. Oh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να συμφωνήσουμε εδώ, σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, για την κοινή αλληλευτική πολιτική των επόμενων χρόνων και μπορούμε να λάβουμε το παράδειγμα του Σκάγερα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το παράδειγμα θα επαναληφθεί. Σήμερα οι αντιπρόσωποι του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Βαλτική βρίσκονται εδώ και χαίρομαι πολύ γι' αυτό και θα ήθελα να τους καλωσορίσω. Πόσο έχει η κατάσταση. Από τη μία μας ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνέχιση της διμερούς συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ορβηγία για την αλληλεία στην περιοχή Σκάγερακ. Από την άλλη, έχουμε και την αλλαγή του κανονισμού για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτά στο μέλλον θα αλλιεύουν με στην περιοχή του Σκάγερακ και με ποιους τεχνικούς ελέγχους και υπό ποιες προϋποθέσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά η Νορβηγία με τις αλλιευτικές πρακτικές της έχει ξεκαθαρίσει ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν είναι και τόσο υποχρεωτική για εκείνους. Τώρα έχουμε συζητήσει εντατικά το θέμα με τους κοιόδης εισηγητές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε ερωτήσεις δικές μου ως εισηγητή αλλά πραγματικά πιστεύω πως πρέπει να συζητήσουμε ουσιαστικά και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ με ερωτήσεις μου στα μέλη του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική. Από ό,τι βλέπω συμφωνείτε. Τώρα, σε γενικές γραμμές, κύριε Κούνλιο Πρόεδρος, ένα λεπτό. Συγγνώμη, θα έπρεπε τον προτέρων να είχα καλωσορίσει στην Επιτροπή μας τα μέλη του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική που βρίσκονται στην αίθουσα είναι φιλοξενούμενοι μας και είναι εν εδώ ακριβώς για να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν ε, ερωτήσεις που θέλετε να απευθύνετε στους εκπροσώπους του Συμβουλίου, ο κύριος Βίτσμαν θα τις απαντήσει εκ μέρους του ΡΑΚ, εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γνωμοτικού Συμβουλίου για την Βαλτική. Συγγνώμη, έπρεπε να το είχα κάνει πριν, αλλά αφαιρέθηκα, λέει ο Πρόεδρος. Το κάνω πάντως τώρα. Λοιπόν, έχοντα διευκρινίσει προς όλα τα μέλη, προσκαλώ τον κύριο Κούν να θέσει τα ερωτήματα που θέλει να απευθύνει στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Και συγκεκριμένα στον κύριο Γουίτσμα, που πρόκειται να απαντήσει και να διευκρινίσει αφιβολίες που υπάρχουν ή να αποσαφηνίσει ερωτήματα. Συγγνώμη, διακοπή κύριε Κούν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Περιφερειακή Επιτροπή για τους επιμέρους από τις επιμέρους περιοχές αποτελείται από εξαιρετικούς εμπειρογνώμονες και αυτό είναι πολύ καλό από συνδέσμους, από ενώσεις αλλιέων, από αντιπρόσωπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και από εθνικές αρχές. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την προετοιμασία του βασικού κανονισμού, ανέφερε διάφορα νούμερα, διάφορους αριθμούς για τις απορρίψεις τα τελευταία χρόνια στους ε, διάφορους ε, αλληλευτικούς ε, τόπους. Περίπου 50-60% των συνολικών αλλιευμάτων αποτελούν αυτές οι απορρίψεις. Δεν ξέρω πώς προέκυψαν αυτά τα νούμερα, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου εάν έχετε εσείς πληροφορίες για το ποσοστό των απορρίψεων στο Σκάγερακ. Για μας επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον αριθμό των σκαφών που αλλιεύουν στην περιοχή. διότι παρότι έχουμε διάφορα συστήματα παρακολούθησης και εντοπισμού που μας λένε ποια σκάφη, με ποια ταχύτητα, σε ποια δρομολόγια λειτουργούν, θα ήθελα εν τούτης να ρωτήσω εσάς. Μετά, όσον αφορά το θέμα του ελέγχου και τις δυνατότητες παρακολούθησης με, ε, κάμερα κλειστού κυκλώματος. Θα ήθελα να ρωτήσω και εκεί τι γίνεται. Μετά, άρθρο 3, υποχρέωση εκφόρτωσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει εξαιρέσεις για, ορισμένους, για ορισμένα αλλιεύματα που έχουν υψηλό ποσοστό επιβίωση σε περίπτωση απόρριψης, για παράδειγμα. Ή για, για μικρούς αλληλείς οι οποίοι δεν ε, αντέχουν οικονομικά να κρατήσουν τα ελλείμματα στο πλοίο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς προκύπτει ο αριθμός, ε, το ποσοστό επιβίωσης των ψαριών, πώς ξεχωρίζεται τα διάφορα είδη, τι γίνεται, ποιες δυνατότητες υπάρχουν εφαρμογής Έχετε αναφέρει κάποια είδη ηχθείων στο τέλος, στο παράρτημα. Και αναφέρετε χρονική προθεσμία το 2014-2015, αν, αν δεν κάνω λάθος. Ε, ερώτηση, πώς κρίνετε εσείς μία πιθανή αύξηση των ΤΑΚ Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη το ποσοστό των απορρίψεων, τη βιομάζα, τα αλλιευτικά αποθέματα και πόσο αυτά μπορούν να πληγούν, την θνησιμότητα των διαφορών ειδών. Χρειαζόμαστε στοιχεία εδώ, επιστημονικά στοιχεία. Μετά, όσον αφορά το συνολικό ποσοστό αλλιεύματος, τι ποσοστό από αυτό το αλίευμα είναι παραλίευμα. Ποιο ποσοστό υπερβαίνει της ποσόστοσης. Ποια κράτη-μέλη μπορούν μέσω ενός συντονιστικού οργάνου να προβλέψουν ενδεχομένως ανταλλαγή ποσοστώσεων. Τώρα, όσον αφορά τα εχθίδια. Έγινε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι καλή, ειδικά, όπου, ειδικά στο σημείο που αναφέρεται η χρήση των ηχθιδίων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. αν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους πίσω στους μήνους από το οποίο λιεύτηκαν. Μετά χρειαζόμαστε πιο ξεκάθαρους ορισμούς για το μέγεθος του ματιού των δικτυών. Μας, λέ... μας αναφέρεται κάποια μέτρα, κάποια χιλιοστά, μας συγχωρείτε. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, τα 35 χιλιοστά για παράδειγμα, για ορισμένους τύπους δικτυών. Όσο εμπειρογνώμονες λοιπόν, ερώτησή μου είναι, θεωρείτε εσείς αυτούς τους αριθμούς Σωστού Και τέλο, τελευταία μου ερώτηση, ηλεκτρονική παρακολούθηση. Ο συνάδελφος Κρίστενσεν, ο σκιώδη εισηγητής, αναφέρθηκε στις πρακτικές της Δανίας, της χώρα του. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν εθελοντικά μέσα ελέγχου, τα οποία συνδέ... Ε, για παράδειγμα με τηλεόραση κλειστού κυκλώματος που συνδέονται με τα ΤΑΚ. Επιπλέον, θα με ενδιαφέρε να μάθω την εμπειρία του Συμβουλίου σχετικά με το πόσο εφαρμόσιμο, εφαρμόσιμη είναι αυτή η τεχνική κλειστού κυκλώματος, ε, τι προβλήματα ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν με την προστασία των δεδομένων και τέλος το ζήτημα της χρηματοδότησης. Ο τεχνικός αυτός εξοπλισμός, οι κάμερες, πάνω στα λιευτικά σκάφη, πόσο θα κοστίσει, προβλέπονται επενδύσεις. Είναι πολύ σημαντικό, τέλος, για εμάς να μάθουμε από εσάς, ως επιρρογνώμονες, την κατάσταση εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά μία παρακολούθηση με τεχνικό εξοπλισμό όλων των αλληλευτικών σκαφών. Εσείς θεωρείτε πως οι αλληλείς και τα σκάφη αυτά μπορούν να το κάνουν. Μπορείτε να τους έχετε εμπιστοσύνη. Κλείνοντας θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω τα μέλη του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και χαίρομαι για την επικοδομητική συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κούν. Θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ε, ευρωβουλευτές και μετά στο ΡΑΚ. Ε, Ευχαριστώ. Με αφορά ιδιαίτερα αυτή η έκθεση. Είναι προφανές ότι θέλουμε να μειώσουμε τις απορρίψεις στο Σκάγερακ. Όμως είναι ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο βιαζόμαστε να προωθήσουμε και μου δημιουργεί κάποια σύγχυση. Ο, υπουργός, ο Δανός υπουργό Τροφίμων ε, είπε ότι οτιδήποτε υιοθετηθεί θα εφαρμοστεί από το 2014 και μετά θα μπορούσε η Κομισιόν να μου το επιβεβαιώσει. Χρειαζόμαστε επίσης ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας σωστά. Θα ήταν καλή ιδέα να περιμένουμε μέχρι το 2014 για να μην κάνουμε λάθος, να μην κάνουμε λάθη. Νομίζω ότι βιαζόμαστε πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές ασάφειες αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να πούμε στους αλληλείς ε, βακαλάου και γάδου στη Βαλτική, το πώς θα αλλιεύουν από 1η Ιανουαρίου και μετά. Ε, θα ήθελα ε, κάποια σχόλια από την Κομισιόν ε, και από το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Οι, οι κανόνε για τα νορβηγικά σκάφη δεν είναι σαφεί, για παράδειγμα. Τα νορβηγικά σκάφη θα πρέπει να αλλιεύουν με του ίδιου όρου που αλλιεύουν και τα ευρωπαϊκά σκάφη. Ε, ε, αυτό συμπεριλαμβάνει και του ε, κανόνε ελέγχου στο Σκάγερακ. Θα μπορούσε η Κομισιόν να μας το διευκρινίσει. Ε, το άρθρο 1 πρέπει να το ερμηνεύσουμε με αυτόν τον τρόπο ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και για τα νορβηγικά σκάφη. Μετά, έχουμε όλο ότι και αυτοί θα έχουν την υποχρέωση ε, να φέρουν κάμερες κλπ. Μετά, στην νομοθεσία ε, θα προβλεφθεί ε, από τώρα, ποια ε, ποια ήδη θα καλυφθούν από την απαγόρευση απορρίψεων ε, στη δεύτερη φάση. Μήπως θα πρέπει να περιμένουμε την ενδιάμεση έκθεση για να το αποφασίσουμε αυτό. Μετά, η Κομισιόν θα διαγράψει την, τον κανόνα για, τα, για την ισχύ ανά ημέρα, τα κιλοβάτα ανά ημέρα. Επίσης, αν γίνει μια εξόρμηση ε, στο Σκάγερακ και στην Βαλτική θάλασσα, όλη αυτή η εξόρμηση, όλο αυτό το ταξίδι θα καλύπτεται από την εξαίρεση από τον κανόνα των απορρίψεων. Ε, από τον κανόνα των κιλοβάτ, συγγνώμη. Μετά, για τα είδη τα οποία καλύπτονται από, την, από την, την απαγόρευση απορρίψεων ε, στη συμφωνία με την Νορβηγία ε, υπάρχει μια ευελιξία 20% ε, του πρώτου έτους, 15% το δεύτερο και 10% το τρίτο. Μήπως θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε καλή, περισσότερη ευελιξία. Σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις τώρα. Οι Υπουργοί Αλίας, Νορβηγίας, Σουηδίας και Δανίας ε, είπαμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η κατανομή των ποσοστώσεων ε, και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη του Περιφερειακού Νομοτικού Συμβουλίου Βόρεια Θάλασσα. Επίσης υπάρχει μια έκφραση για στο, στο έγγραφο για την αύξηση της περιφερειοποίησης. Θα ήθελα όμως να μην βιαστούμε πάρα πολύ, να είμαστε σίγουροι για το κείμενο το οποίο θα εγκρίνουμε έτσι ώστε να λειτουργεί αντί να δημιουργεί απογοητεύσει και προβλήματα. Ευχαριστώ. Κύριε Λέβιν. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τον κύριο Κούν ω συζητητή. και καλωσορίζουμε και όλου του εμπειρογνώμονε από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο τη Βαλτική. Χαίρομαστε πολύ που σα έχουμε για να συζητήσουμε δύο πράγματα. Καταρχά, συμφωνώ απολύτω με τον ε, κύριο Κρίστενσεν ότι αισθανόμαστε κάπως δεγμένοι ε, συζητώντας αυτά τα θέματα. Με δεδομένο ότι ο Δανός Υπουργό Διατροφέ είπε ότι θέλει μια, ένα προσχέδιο να αποσύρει την πρότασή τη. Η Επιτροπή δεν έχει αποσύρει την πρότασή τη, άρα πρέπει να συνεχίσουμε το δουλειά μα εδώ. Το ερώτημα όμω είναι τι θα κυριαρχήσει. Ο κύριος Κούντ θα πρέπει να καταλήξει πώς θα λειτουργήσουμε. Και αναρωτιέμαι, γιατί τι σκέφτεται ο Δανός υπουργό. Το ερώτημα ήταν ότι υποτίθεται έπρεπε να έχουμε αυτή την ε, απαγόρευση ε, ε, ε, ανεξαρτήτως των ε, ποστών που θα τεθούν. Και ελπίζω από το 2014 να έχουμε μια νέα κοινή αλλιευτική πολιτική, βασικό κανονισμό δηλαδή, με μία μόνο απαγόρευση για τις απορρίψεις, σε κάποια μορφή. αυτή η πρόταση τότε αυτόματα θα είναι επιχειωμένη και θα απορριφθεί. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη τη επιτροπή επί του θέματος. Αλλά θα ήθελα επίσης και δεδομένη την ευκαιρία ότι έχουμε τους εμπειρογνώμονες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Βαλτική, να ακούσουμε και τη δική του άποψη για το πώς θα έπρεπε να είναι και πώς πρέπει να διαμορφωθεί η πρόταση αυτή. Κάποιε ερωτήσει που θα ήθελα να θέσω. πρέπει να λειτουργήσουμε αυτά τα ελάχιστα μέτρα που δίνονται στο παράρτημα της ε, πρότασης. Δεν είναι το ελάχιστο ε, ε, για το ελάχιστο σε ό,τι αφορά τα μάτια των δικτυών, αλλά το ελάχιστο, ε, συγγνώμη, δεν είναι το θέμα του ελάχιστον εκφορτώσεων, αλλά ε, η ποσότητα Εάν δούμε τα ελάχιστα μέτρα για τον Βακαλάο, είναι 32, 33 έως 35 ε, ε, μιλιμέτρ, που είναι εξαιρετικά μικρό, ε, εκατοστά, συγγνώμη, που είναι ουσιαστικά δεν είναι καθόλου ενδιαφέρον εμπορικά μέγεθος. Αναφέρομαι λοιπόν, προς, στον κύριο Χέντρισον, που είναι από, την, από το Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, και οι Σουηδοί θέλουν ότι θέλουν πολύ υψηλότερο ε, ελάχιστο μέγεθος για το επιτρεπόμενο αλίευμα. Θέλουμε βέβαια να αποφύγουμε στο δυνατόν είδη τα οποία δεν είναι βιώσιμα εμπορικά για να έχουμε λιγότερες απορρίψεις. Άρα θα πρέπει ίσως να αυξήσουμε το μέγεθος τον, ε, το κατόφλι το οποίο έχει τεθεί για το αλλιευόμενο είδος. Και στην πράξη όταν ε, κατονομίζουμε, κατονομάζουμε αυτή τη σειρά ειδών, όπως το κάνουμε στο παράρτημα, τι θα σκεφτούν σχετικά οι αλληλείς. Είναι πρακτικά εφικτό για αυτούς να έχουμε όλο αυτό τον κατάλογο και να απορρίπτουμε, αν θέλουμε, όλο αυτό τον κατάλογο ε, ειδών που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στι απορρίψει. Υπάρχουν και πολλά πολλά περισσότερα είδη. Είναι ατελείωτο ο κατάλογο. Άρα δεν είναι πρακτικό να συμπεριλαμβάνεται ένα κατάλογο. σω το απλούστερο θα είναι ακριβώ ότι να, έχεις, ε, να επιβάλλεται μεγαλύτερο μέγεθο ματιών στα δίκτυα για να, αποφυγούν, για να αποφευχθούν υπερβολικά πολλέ απορρίψει ε, ε, Και επομένω τελικά έχοντα το μεγαλύτερο αυτό μάτι, ουσιαστικά αυτό το οποίο αλλιεύεις είναι αυτό το οποίο σου επιτρέπεται να εκφορτώσεις. Άρα, το επόμενο ερώτημα που ερχόμαστε. Το παράδειγμα το οποίο αφορά στα είδη. Δεν θα ήταν καλύτερο να συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη, αλλά με πολύ, σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, επιτρεπόμενο μέγεθος αλλιεύση. Και στη συνέχεια, το κλειστό κύκλωμα τηλεόραση και την παρακολούθηση. Δεν υπάρχει σε πολλά κράτη και προτείνεται εδώ να το έχουμε εμείς. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η Νορβηγία ισχύει το σύστημα αυτό πριν από 30 χρόνια, όταν δεν είχαμε τέτοιου είδου εμεί συστήματα, το κύκλωμα ε, κλειστή τηλεόραση, την παρακολούθηση. Τώρα ξέρω βέβαια ότι ναι, μεν η Νορβηγία δεν είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και πολύ καλό παρελθόν σε ό,τι αφορά την αλίευση στα νορβηγικά ύδατα ή και απόρριψη σε ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, σε χωρικά ύδατα τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα αλλιεύματα τα οποία δεν επιτρέπονται. Άρα καταλαβαίνουμε τον προβληματισμό τη ναυπηγίας από του θέματο και θα πρέπει να φύγουμε από αυτή την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν. Και ευχαριστώ περιμένουμε και προσβλέπουμε να ακούσουμε τι απόψει των ορδηγών αλλιέων που μπορεί να είναι πάρα πολύ επικοδομητική ακριβώς ε, η πρόταση. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέλω να αποβάλω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλώς ορίζουμε τον κύριο Βίτμαν και του δίνουμε το λόγο για να απαντήσει τα ερωτήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια καταρχήν. Είμαι ο Νίλ Σβέκμαν, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Νομοτικού Συμβουλίου Βόρειας Θάλασσας. Εργάζομαι στην ε, Δανέζικη Ένωση ε, Αλλιεών. Δίπλα μου έχω τον πρόεδρο της οργάνωσης αυτής και πιο πέρα ο κύριος Άντερσον είναι ε, ο πρόεδρος της ε, είναι επίση εκτελεστικό μέλος του, του, είναι μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του ΡΑΚ και πιο δίπλα ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας του ΡΑΚ της Βόρειας Θάλασσας που ε, ασχολείται με ζητήματα του Σκάγερα και του Κάτεγατ. Έχω και κάποιους χάρτες πώς μπορείτε να τους ε, διανύμετε στα μέλη της Επιτροπής που δείχνουν που βρίσκεται το Σκάγερακ. και ποια είναι η οριοθέτηση ανάμεσα στο Σκάγερα και τη Βόρεια Θάλασσα, όπως επίσης και ανάμεσα στο Σκάγερα και το Κάτεγατ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γεωγραφικά για ποια περιοχή μιλάμε. Είναι μια περιοχή που σχετίζεται στενά με τις άλλες δύο, το Κάτεγατ και τη Βόρεια Θάλασσα. Και υπάρχουν και κάποια νούμερα σε, που είναι η καταπροσέγγιση, το καταπροσέγγιση όγκος των αλλιευμάτων για τους δανούς αλλιείς. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια συμφωνία Σουηδίας, Νορβηγίας και Δανίας ανάμεσα βασικά στους Υπουργούς Αλίας και την Ταμανάκη. Ε, που υποστήριξαν την πρωτοβουλία για την απαγόρευση απορρίψεων. Αυτό αποτελούσε τμήμα της συμφωνίας με την Νορβηγία, του συμφωνητικού με την Νορβηγία του 2011. Αυτό οδήγησε και στην απαγόρευση της 4ης Ιουλίου. Η Κομισιόν υπέβαλε την πρότασή της στις 29 Αυγούστου ε, και εμείς τελούμε από την ίδια σύγχυση που τελούν και όλοι οι υπόλοιποι. Ο υπουργό Δανίου, ε, Δανίας ε, είπε ότι ε, η υπαγόρευση αυτή μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή και μάλλον μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μετά το 2014. Όμως δεν μας ζητήθηκε η γνώμη. Δεν μας ζητήθηκε η γνώμη στο ΡΑΚ Βόρειας Θάλασσας. Υπάρχει παρόλα αυτά μια ομάδα εργασία που παρακολουθεί την, κανονικά τις ε, διαπραγματεύσεις με την Νορβηγία. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα της διαπραγμάτευσης με την Νορβηγία. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κανονός είδους μελέτη αντικτύπου αυτής της πρότασης. Φαντάζομαι ότι αυτό συνέβη επειδή βιαζόντουσαν. Ε, σε τέτοιου είδους όμως περιπτώσεις, αν κανείς αναρωτιέται αν το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Διαρωτώ με ποιος έχει δικαιώματα, αλληλευτικά δικαιώματα εκεί. Είναι και η Γερμανία, είναι το Βέλγιο, είναι και οι κάτω χώρες που έχουν αλληλευτικά δικαιώματα. Δεν είναι μόνο η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία. Η Γαλλία επίση και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν ποσοστότηση, αλλά έχουν δικαίωμα κάποια αλίευση και στο Σκάγερακ, γιατί για ορισμένα είδη έχουν το δικαίωμα να αλλιεύουν είτε στη Βόρεια Θάλασσα είτε στο Σκάγερακ, Όπω επιθυμούν. Συνεπώ έχουμε 7 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπλέκονται. Δεν είναι μόνο ζήτημα ε, των σκανδιναβικών χωρών, ούτε μόνο τη Δανία. Παρόλο ότι βέβαια η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία έχουν τα περισσότερα αλληλευτικά δικαιώματα. Το συζητήσαμε στο Περιφερειακό Γνωματικό Συμβούλιο της Βόρειας Θάλασσας και είπαμε ότι ενδεχομένως η απαγόρευση απορρίψεων να είναι η σωστή λύση. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι, το γεγονό ότι ελήφθη πολιτική απόφαση μα υποχρεώνει να δούμε πώ μπορούμε να χειριστούμε προ το καλύτερο όφελο των αλλιών μα το ζήτημα αυτό. Οπότε πρέπει να δούμε ποιε είναι οι διευκρινήσει που ζητούμε. Ε, θα τα επαριθμίσω όλα αυτά τα θέματα τα οποία μα απασχόλησαν και ενδεχομένω θα απαντήσω και σε ορισμένε ερωτήσει που έγιναν. Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί αυτή η απαγόρευση απορρίψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε καλό είναι να τα κάνουμε σωστά τα πράγματα και όχι γρήγορα. Οπότε, γιατί αυτά τα 15 είδη και όχι όλα. Πολύ καλή ερώτηση. Και αυτό δεν το έχουμε συζητήσει επαρκώς. Ποιο είναι το κριτήριο με βάση το οποίο καθορίστηκαν αυτά τα είδη. Ίσως το γεγονός ότι οι ποσοστώσεις με για αυτά τα είδη συμπληρώνονται πιο γρήγορα. Αν για παράδειγμα έχω καλύψει την ποσόστοσή μου τον Απρίλιο, τι πρέπει να σταματήσω να αλλιεύω για το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο χρόνο. Στην Σουηδία ε, απαγόρευσαν τον Αύγουστο την περαιτέρω αλλιεύση γάδου. Ε, και με την απαγόρευση απόρριψης ε, οι αλληλείς θα πρέπει να σταματήσουν να αλλιεύουν τελείως. Αυτό θα πρέπει να το λύσουμε. Δεν θα πρέπει να έχουμε ειδικού όρους για τα σκάφη έτσι ώστε να μπορούν να διατηρούν τα προς απόρριψη αλλιεύματα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους. Δεν θέλουμε να απορρίπτουμε γιατί τα ψάρια που μπορούν να καταναλωθούν θα πρέπει να εκφορτώνονται και όχι να απορρίπτονται. Αλλά μετά λέγεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά για αναπτυξιακή βοήθεια, για ζώα συντροφιάς ε, κλπ. Αλλά ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι η αναπτυξιακή βοήθεια που περιλαμβάνει ψάρι ε, δεν είναι επιτυχής, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να φάνε ψάρι. Μετά, γιατί χρειαζόμαστε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς. Όσο μεγαλύτερο είναι το ψάρι, τόσο πιο πολύτιμο είναι. Αυτό είναι γεγονός. Και ασφαλώς οι αλληλείς θέλουν να βελτιστοποιήσουν την αξία των ελευμάτων τους. Συνεπώ, κανεί δεν θα θέλει να ε, ψαρεύει και ένα πολύ ε, ηχθίδια. Πόσο ψηλό θα πρέπει να είναι το πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το μέγεθος ε, εξαρτάται. Μπορούμε να ζητήσουμε τη γνώμη του Άισες για να δούμε τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι ποσοστώσεις ε, τις οποίες καθορίζουμε. Η Κομισιόν δεν έχει α, απευθύνει στην ISIS. Έχουμε την εντύπωση ότι για ορισμένα είδη οι είναι πιο ψηλές από ότι για άλλα. Ε, αντιθέτως όμως θα πρέπει να διατηρήσουμε την ίδια θνησιμότητα για όλα τα είδη. Όμως θα πρέπει να καθοριστούν οι αρχές. Θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση. Έχουμε κοινέ ποσοστώσει επίση για τη Βόρεια Θάλασσα και το Σκάγερακ. Πώ θα τι κατανείμουμε, Αν για το Σκάγερακ εφαρμόζεται ένα ιδιαίτερο σύστημα, τα ψάρια δεν γνωρίζουν σύνορα. Εμεί έχουμε όμω ποσοστώσει κοινέ για Σκάγερακ και κάτεγατε επίση. Τι, θα έχουμε ένα σύστημα για το Σκάγερακ που δεν ισχύει για τις άλλες περιοχές. Και πώ θα εξασφαλίσουμε για την ετήσια ευελιξία. Και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ευελιξία θα είναι προς όφελος των σκαφών. Γίνεται λόγο επίσης για πλήρη τεκμηρίωση, για παρακολούθηση από ε, τηλεόραση κλειστού κυκλώματος κλπ. Δεν είναι μυστικό ότι οι αλληλείς, στους αλληλείς δεν αρέσουν αυτά τα συστήματα, αλλά αν είναι να επιλέξουμε αυτά τα συστήματα θα πρέπει να δούμε με ποιους όρους θα χρησιμοποιούνται. Και μετά πρέπει να δούμε ε, οι τρεις βόρειες χώρες ε, έχουν 600 σκάφη συνολικά που αλλιεύουν εκεί. Αν είναι να εγκαταστήσουμε συστήματα κλειστού κυκλώματος σε όλα αυτά τα σκάφη, αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να επίσης τίθενται και άλλα θέματα. Σε ποιον ανήκει το οπτικό υλικό. πόσο καιρό θα πρέπει να, διατηρούν, να διατηρείται αυτό το υλικό. Και μετά, ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Δεν είναι τον όλοι να έχουν πρόσβαση. Κατόπιν, ε, το θέμα των, ε, της, ε, του κανονισμού αλληλευτικής προσπάθειας. Αν χρειάζεται πλήρης τεκμηρίωση, αυτό σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να το να δούμε και τον κανονισμό αλληλευτικής προσπάθειας. Μετά, για τους ελέγχους. Μπορούν να γίνουν πλήρης έλεγχοι. Ο πλήρης έλεγχος δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται μέσω κάμερας. Η Νορβηγία δεν πιστεύει σε τέτοιου ε, κάμερες για μας, για την Ορβηγία μάλλον, πλήρης έλεγχος είναι ε, οι επιθεωρητές στο σκάφος κλπ. Τι γίνεται όταν τα αλλιευτικά σκάφη αλλιεύουν σε διάφορες περιοχές, κάτι που σημαίνει πολύ συχνά στη Βόρεια Θάλασσα, το Σκάγερα και το Κάτεγατ. Τι γίνεται με τους ελέγχους σε αυτή την περίπτωση. Και μετά, θα έχουμε διαφορετικούς κανόνες ελέγχου για τα σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφορετικούς για την Νορβηγία, γιατί οι Νορβηγοί δεν δέχονται τις κάμερες. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα αλλιεύουν στα νερά αυτά χωρίς κάμερες και εμείς αντίστοιχα θα κλείνουμε τις κάμερές μας στα νορβηγικά ύδατα. Όχι βέβαια, οπότε τι, θα εφαρμόζονται δύο διαφορετικοί κανόνε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των αποθεμάτων και την επιστημονική γνώμη. Όταν αποκτήσουμε σύστημα με ποσοστό σαλευμάτων και πρέπει όλα να εκφορτώνονται, τότε θα αντιμετωπίσουμε σοβαρότατα προβλήματα με τις καθυστερήσεις στις επιστημονικές νομοδοτήσεις. Θα σας δώσω το εξής παραδείγμα έχουμε διάφορα είδη των οποίων τα αποθέματα αυξάνονται. Ένα παράδειγμα είναι ο μπακαλιάρο στη Βόρεια Θάλασσα, στο Σκάιρα και το Κάτεγατ. Οι επιστημονικές νομοθετήσει όμως έφτασαν πολύ καθυστερημένα και τι είχαμε κάνει, είχαμε μειώσει την αλληλευτική μας προσπάθεια ήδη. Οπότε θα θέλαμε να μπορούμε να συνεχίσουμε την αλίευση. Και να μην λαμβάνουμε απότομα και κατεπήγοντα μέτρα. Θα πρέπει η παρακολούθηση, η επιστημονική παρακολούθηση να είναι πραγματικού χρόνου, γιατί αλλιώς τα πράγματα δυσκολεύουν. Οπότε εκεί το θέμα μηχανισμού λήψης αποφάσεων. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια περιφερειακή προσέγγιση για την διαχείριση σε καθημερινό επίπεδο των αλλιευμάτων. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στον, στα διάφορα ΡΑΚ, την ε, Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Και σίγουρα εδώ χρειάζονται ε, πράξεις κατεξιοδότηση. Αυτές είναι ορισμένες από τις ερωτήσεις. Λίγες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση και για το γεγονό ότι δεν μας παρουσιάσετε όλες τις ερωτήσεις. Η Κομισιόν θέλει το λόγο. Yes, thank you, and apologies that I was a little bit... Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που άργησα κάπως. Θα αρχίσω με αυτό που άκουσα όταν μπήκα για τις αυξήσεις στα ΤΑΚ. Αληθεύει πως εάν πρέπει να προσμετρούμε όλα τα αλλιεύματα για τις ποσοστώσεις πρέπει να, και να εκφορτώσουμε δηλαδή όλα τα αλλιεύματα, οι ποσοστώσεις πρέπει να αυξηθούν. Έχουμε στείλει ένα αίτημα στο ISIS. Όμως μας απάντησαν το εξή. Επειδή δεν έχουν ξεχωριστές πληροφορίες για το Σκάιερα και τη Βόρεια Θάλασσα, θα χρειαστούν να αντιμετωπίσουν ξεχωριστά το θέμα αυτό και θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να απαντήσουν στο αίτημά μας. Υπάρχει λοιπόν μια καθυστέρηση σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, αλλά αναγνωρίζουμε πως υπάρχει ανάγκη τα νούμερα να είναι σωστά, γιατί αυτό που δεν θέλουμε είναι να μην αφήσουμε ελαστικά περιθώρια για αυτή την απαγόρευση των απορρίψεων και είχαμε ήδη άσχημες εμπειρίες από την πρώτη εφαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν επιθυμούμε να έχουμε τα σωστά στοιχεία πρώτου προχωρήσουμε από το ISIS για να μπορέσουν οι αλείς να συνεχίσουν και η αλία να είναι πιο κερδοφόρα, διότι από τη στιγμή που εκφορτώνεις το αλίευμα θα πρέπει και να είσαι στην θέση να αυξήσεις την αξία του. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο να το πετύχουμε αυτό τον πρώτο χρόνο. Θα προσπαθήσουμε όμως, όσο μπορούμε. Τώρα, αναφέρθηκε το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης. Αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρουμε λαμβάνοντας υπόψη και τις συζητήσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα όσον αφορά είδη ψαριών που έχουν μικρότερο μέγεθος από το επιτρεπόμενο. Για το σκάγερα και ισχύουν και αυτά που έχουμε πει στην πρόταση μεταρρύθμισης, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα ψάρια που έχουν μέγεθος κάτω από το επιτρεπόμενο για ανθρώπινη κατανάλωση και για να το εφαρμόσουμε χρειαζόμαστε την τήρηση του ελάχιστου μεγέθους. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αγορά για αυτά τα μικρά ψάρια. Αυτό βέβαια είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Νορβηγοί, δηλαδή να πουλήσουμε όλο το αλίευμα, όλη την ψαριά ή όχι. Αλλά να μην, έχουμε, να μην απαιτήσουμε την ίδια τιμή για τα ψάρια που έχουν μικρότερο μέγεθος, για τα ηχθίδια. αυτή τη στιγμή ο κανονισμός ε, για το Σκάγερακ αντανακλά αυτά που έχουμε ήδη συζητήσει και αυτό περιλαμβάνονται στον κανονισμό. Τώρα, αναφέρθηκε το ερώτημα του τι γίνεται με, το, με τον μπακαλιάρο, για παράδειγμα, για τα αποθέματα μπακαλιάρου στη Βόρεια Θάλασσα και στο Σκάγερα και τις επικαλύψεις βασιζόμενοι στις εκτιμήσεις που έχουμε για τα ποσοστά απορρίψεων στο Σκάγερακ θα χρειαστεί αύξηση των ΤΑΚ. Αλλά θα χρειαστούμε κάποιες ρήτρε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα λεύματα αυτά δεν θα ε- εξαχθούν προς τη Βόρεια Θάλασσα. Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Δεν σας λέω ότι είναι εύκολο. Και υπάρχει κάτι που είναι ακόμα πιο περίπλοκο με τις αυξήσεις, με το Σκάγερακ, με την Βόρεια Θάλασσα, ότι πολλά από τα αποθέματα τα μοιραζόμαστε με την Νορβηγία. Και αυτά τα για αυτά τα αποθέματα πρέπει να συμφωνήσουμε με τους Νορβηγούς για το ποσοστό των ΤΑΚ. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν αυτό το μήνα με την ορβηγία αλλά δεν μπορώ να σας εγγυηθώ για το αποτέλεσμα. Τώρα υπάρχει επίσης μία σάφια για το πότε θα τεθεί σε ισχύ. Θα σας πω λοιπόν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2013 θα τεθεί σε ισχύ. Ο στόχος όμως αυτός είναι πολύ δύσκολος να επιτευχθεί. Ακριβώς γιατί η ISIS δεν μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και θα χρειαστεί 6 μήνες όπως σας είπα. Στόχος μας όμως προς το παρόν παραμένει 1η Ιανουαρίου του 2013. Τώρα το πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Τώρα, δίνουμε ένα χρόνο περιθώριο για τα σκάφη με έως 15 μέτρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 για να εξοπλιστούν με τις κάμερες αυτές και για τα σκάφη με πάνω από τα 12 μέτρα, από 12 έως 15 έχουν έναν επιπλέον χρόνο περιθώριο. Επίσης, πιστεύω πως υπήρξε μια σάφια για τα νορβηγικά σκάφη. Η απαγόρευση απορρίψεων είναι κάτι που έχει συμφωνηθεί με την Νορβηγία. Δεν είναι πανομοιότυπη όμως αυτή η συμφωνία με τις ε, υπόλοιπες απαγορεύσεις απορρίψεων. Συμφωνήσαμε σε κάποιους κοινού κανόνες, κάποιες τεχνικές προδιαγραφές. Η Νορβηγία θα συμμορφωθεί με τα τεχνικά μέτρα αυτά στο Skyerack, θα σεβαστεί την απαγόρευση των απορρίψεων, αλλά η απαγόρευση των απορρίψεων είναι διαφορετική από την νορβηγική απαγόρευση των απορρίψεων και να σας το εξηγήσω κάπως. Η Νορβηγία αφήνει περιθώριο στους αλληλείς να αποφασίσουν αν θα απορρίψουν ή όχι τα αλλιεύματά τους. Δηλαδή, ο ψαράς αποφασίζει αν το ψάρι θα επιβιώσει αν το ρίξει πίσω στη θάλασσα. Αυτό δεν μας άρεσε. Θα θέλαμε σαφέστερους κανόνες Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν ένα από τα είδη ψαριών ε, στο παράρτημα ε, πιαστεί στα δίχτυα σας, πρέπει να το εκφορτώσετε, εκτός από τις εξαιρέσεις τις οποίες μπορούμε να εισαγάγουμε, όπως για τα ψάρια που πιάνονται σε... κιούρτους και κοφινέλα. Νορβηγία όμως θα σεβαστεί τους κανόνες, τους κοινού κανόνες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα τομέα στον οποίο δεν έχουμε συμφωνήσει, στα μέτρα ελέγχου. Έχουμε συμφωνήσει σε κάποια γενικότερα μέτρα ελέγχου στο Σκάγερακ, δεν συμφωνήσαμε όμω σε συγκεκριμένα μέτρα επιβολής απαγόρευσης των απορρίψεων στο Σκάγερακ. Δυστυχώς. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε τις μεθόδους ελέγχου και εποπτείας. Νομίζω πως απάντησα στις ερωτήσεις που άκουσα, αλλά πείτε μόνο, ξέχασα κάτι. Ευχαριστώ. Κυρία Φράγα. Κυρία Φράγα, έχω μια ερώτηση σε σχέση με αυτά που είπε η Κομισιόν. Είπε ότι προτίθεται να αυξήσει τα ΤΑΚ για να αντισταθμίσει την υποχρέωση ε, εκφόρτωσης και λέει ότι αυτό συμπίπτει με το πνεύμα της αναθεώρησης. <laughs> Δεν ξέρω με το πνεύμα, αλλά με το γράμμα σίγουρα δεν συμφωνεί, δεν συνάδει. Νομίζω ότι η Κομισιόν έχει αλλάξει στάση. Γιατί μέχρι τώρα πάντοτε έλεγε ότι η, εκφόρτωση, η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν σήμαινε αύξηση των ποσοστώσεων. Ε, των... Ε, και αυτό είναι κάτι καινούριο, μπορεί να μου το βεβαιώσει η Κομισιόν. Λοιπόν, Μάλιστα, ως εισηγητή στο τέλος θα ήθελα να κάνω μια περίληψη, οπότε νομίζω πως θα ήταν καλό να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Αν θέλετε να το αφήσουμε για το τέλος, ε, γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Αν θέλετε, με, κάνετε τη σύνοψη στο τέλος. Ο κ. Κρίστενσεν. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν, Ευχαριστώ. Η, κυρία, η Επιτροπή λέει ότι η Ευρωβουλία έχει πει ναι να συμφωνήσει στους ίδιους κανόνες, αλλά ταυτόχρονα η Επιτροπή λέει ότι εάν δούμε τα μέτρα ελέγχου και την εφαρμογή τους, τότε κάθε χώρα θα χρησιμοποιήσει τη δική της μέθοδο. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχουμε κάμερες παρακολούθησης πάνω στα νορβηγικά σκάφη. Τότε θα ήταν σαφέστερα τα πράγματα. Εάν δούμε την ημερομηνία που θα δεθεί σε ισχύ ε, η πρόταση αυτή, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξαιρετικά σαφής. Και αυτές οι ασαφείς δηλώσεις μπορούν να προκαλέσουν ευρικότητα ως το τι ακριβώς θα συμβεί όταν δεν ξέρεις πότε θα τεθούν σε ισχύ οι κανόνες. Και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος όταν ε, ο Υπουργό Αλλία μια χώρα λέει ότι θα κάνουμε αναπολύ μέχρι το 2014 και η Επιτροπή λέει ότι θα προσπαθήσουμε να τα θέσουμε όλα σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ακόμα και αν δεν έχουμε έτοιμα τα στοιχεία και τις, ε, τα συγκεκριμένα αριθμιστικά στοιχεία, τότε πραγματικά δημιουργείται τεράστια σύγχυση και είναι εξαιρετικά ευάλωτη βιομηχανία. Θα πρέπει να προετοιμάσω τα πάντα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 ή θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2013 η ημερομηνία ισχύω. Τους είναι αδύνατο να δουλέψουμε αυτές τις συνθήκες. Η απόφασή μας λοιπόν μπορεί να είναι εξαιρετικά κοντόφθαλμη εάν πιέσουμε να υιοθετηθεί η πρόταση αντί να την συντάξουμε με πολύ πιο λογικό τρόπο, όπως λέει το Γνωμονικό Συμβούλιο. Δεν είναι αρκετά σαφής η Επιτροπή του θέματος. Ευχαριστούμε κύριε Τόμας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι στην πράξη περνάμε λίγο τις μεγάλες αρχές, τις μεγάλες θεωρίες, περνάμε στην πράξη και το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλές, ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πολλές θεματικές, παρακάπτοντας τα θέματα αρχής. Καταρχάς, το ζήτημα των ελέγχων και η σημασία εναρμόνισης Εάν θέλουμε πραγματική μεταρρύθμιση και οι τροποποιώσεις αυτές να μην προκαλέσουν σύγκριση και να μην προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα, είναι απαραίτητο όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα αυτό, όλοι οι επαγγελματίε οι οποίοι λειτουργούν στην ίδια ζώνη και σε αντίστοιχα και ίδια αλληλευτικά σκάφη να υπόκειται του ίδιους κανόνες. Διαφορετικά βρισκόμαστε εκ προημίου ε, απέναντι σε προβλήματα και δυνάμει διενέξει και συγκρούσεις. Και οι εξηγήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τελικά ήταν ακόμα πιο ανισχυτικές από ό,τι περίμενα. Γιατί ουσιαστικά τελικά φαίνεται ότι ο ενιαίος κανόνας δεν ισχύει για τους άλλους. Δεν είναι ο ίδιος και ενιαίος κανόνας ότι αφορά τις απορρίψεις και από τη μία το αφήνουμε στη διακριτική ευχέρεια του ψαρά για ένα είδος ένα σε άλλο όχι. Δεν είναι ίδιος ο κανόνα σε ό,τι αφορά τι κάμερε ε, κλειστού κυκλώματο παρακολούθηση, Άρα πάλι υπάρχει κίνδυνο να μην ισχύει ενιαίο ίδιο κανόνα για του πάντε. Δεύτερο πρόβλημα, αυτό των, ε, μέτρη, ε, των ε, μέγιστων επιτρεπόμενων αλλιευμάτων, των τάκ δηλαδή και των απορρίψεων. Ε, Συμμερίσουμε αυτό που είπε ο κ. Κρίστα σε ό,τι αφορά το θέμα τη ημερομηνία και αν δούμε πώ θα, διαμα... θα διαδραματίζονται τα πράγματα και πώ θα εξελίσσονται, ουσιαστικά παρά τις διάφορες διαβεβαιώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει ουσιαστικά κάποια ε, απόλυτη, ε, κάποια συνέχεια αν θέλετε σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή, τη νέα ΚΑΠ και την εφαρμογή της πρότασης αυτής. Εάν δούμε τις, και σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα για τις απορρίψεις, για μένα το, το σημαντικό είναι να είναι βιώσιμη η και η βέλτιστη δυνατή απόδοση. Άρα ο κανόνας ο οποίος θα αφορά στον καθορισμό τις ε, ποσοστώσεις ήταν αυτός που ίσχυε και ξαφνικά ο ορισμός αυτός ε, εξαφανίζεται έναντι των αυτών που δίνονται τώρα και προβλέπονται σε ό,τι αφορά τις ε, απορρίψεις. Άρα πολύ σωστά είπε ο εμπειρογνώμων του ΡΑΚ, εάν θέλουμε οι απορρίψεις αυτές να γίνονται σωστά θα πρέπει να υπάρχουν είτε τα μέσα τα σωστά είτε να δοθούν οι ανάλογες ποσοστώσεις. Οπότε θα πρέπει να δώσουν περισσότερο χρόνο. Κατ' εμέ νομίζω ότι είναι πολύ πιο σόφρο να υπάρχει ένας σχεδιασμός χρονικός, του χρονικού ορίζοντα, συναρτήσει του τι μπορεί να γίνει όντω, του τι είναι εφικτό, συναρτήσει όντω και του μεγέθους και της θνησιμότητα κάποιων ε, ειδών και του βαθμού θνησιμότητα των απορρίψεων και επίσης ελέγχθη κατά κόρον στην Επιτροπή αυτή τα αλλιεύματα δεν ε, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ε, σε ό,τι αφορά τις ε, απορρίψεις και εκεί δεν είναι σε αυτά τα πράγματα. Το κατακλείδι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στην ε, όλη συζήτηση και θα το βρούμε και σε άλλες συμφωνίες το ζήτημα της αντιμετώπισης του θέματος αναπεριφέρεια. Το συζητήσαμε, το είδαμε ήδη στον ελληνικό το θέμα ακριβώ τη αντιμέτωπη των θεμάτων αναπεριφέρεια είναι σημαντικό γιατί επιτρέπει εναρμόνιση των ελέγχων, των προσεγγίσεων, επιτρέπει στι ε, διαφορετικά ληφτικά σκάφη να, να αλλιεύουν στην ίδια ζώνη με ίδιου και κοινού κανόνε που θα είναι αποτελεσματικοί. Γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα αναγεωγραφική ζώνη. Και πραγματικά εκπλήττομαι και θα ήθελα να έχω την αντίδραση επιτροπή του θέματος Εάν δεν υπήρξε διαβούλευση των προτέρων με το γνωμοδοτικό συμβούλιο πάνω στο θέμα αυτό, πραγματικά προξενεί κατάπληξη και είναι αρνητικό στοιχείο. Και για το μέλλον δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Ρόντουστ. Και... Μάλιστα, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο Τόμας. Και ως υπεύθυνη για τον κανονισμό μπορώ να πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένη. Διότι όπως διαβάσαμε στην πρόταση της Κομισιόν, η απαγόρευση των απορρίψεων πρέπει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν συντομότερα, εάν γίνεται από την 1η του 2013 για όλα τα είδη. Ελπίζω να εφαρμοστεί και να συμπεριληφθεί, στον, να συμπεριληφθεί μάλλον στον κανονισμό για το Σκάγερα, γιατί για μένα είναι κάπως σαν πιλωτικό project αυτό και ίσως δεν έχω καταλάβει καλά, αλλά από ό,τι ακούω, η συνεργασία ανάμεσα ε, στο Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβόλιο και στην Κομισιόν δεν είναι καλή και λυπάμαι γι' αυτό. Άκουσα ότι τα στοιχεία είναι αόριστα, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι όντως θα εφαρμοστεί από 1η Πρώτου 13 δεν υπάρχει κάποια καλή ρύθμιση για τα μεταναστευτικά είδη, δεν υπάρχει κάποια σαφής ρύθμιση για τα μέτρα ελέγχου. Όπως είπατε η Νορβηγία ελέγχει μόνη της τα δικά της σκάφη, άλλες χώρες μόνες τους τα δικά τους. Υπάρχει γενικότερη ασάφεια στους ελέγχους και να πραγματικά Είμαι πολύ σκεπτική με όλα αυτά που άκουσα και σας παρακαλώ να μου απαντήσετε τι θα κάνουμε με το βασικό κανονισμό. Εάν έχουμε προβλήματα ήδη τώρα που κάνουμε κάτι πιλωτικά, τι θα γίνει στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Κύριε Μάλιστα. Και εγώ συμφωνώ με την κυρία ότι Είμαι πολύ απογοητευμένη με τις εξελίξεις και με το πώς ε, διεξήχθησαν όλα αυτά. Υπήρχε ένα θετικό πνεύμα ε, το 2011 στους τρεις μεταξύ των τριών υπουργών Αλίας και τώρα τι γίνεται. Τώρα υπάρχουν καθυστερήσεις. Κανείς δεν συμβουλεύετε τους ε, υπολείπους. Εμείς εδώ ως κοινοβούλιο το μαθαίνουμε στο τέλος. Πού έγινε λάθος, πείτε μου. Μήπως υπάρχει έλλειψη πολιτικής θέλησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήλπιζα με αυτή, ε, αυτή η πρόταση να είχε παρουσιαστεί νωρίτερα εδώ στο Κοινοβούλιο Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό που μας είπατε για την 1η Πρώτου 13, τι περιμένετε. Ποιες αποφάσεις περιμένετε, τι θα σας επηρεάσει για να αλλάξετε κάτι και τι περιμένετε από εμάς. τίποτα δεν είναι σαφές. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε την ε, μεταρρύθμιση και να απαγορεύσουμε τις απορρίψεις, μας κάνετε πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να ήθελα να σχολιάσω όσα είπε ο κύριος Βίκμαν ως πρόεδρος του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική. Αναφέρθηκε το ελάχιστο μέγεθος για τη διατήρηση των πληθυσμών. Τώρα, για τα ηχθίδια. Δεν θα έπρεπε να εισαγάγουμε και εκεί ελάχιστο μέγεθος. Γι' αυτό πιστεύω πως θα έπρεπε να πείτε ότι πρέπει να αυξηθεί το μέγεθος ματιών στα δίχτυα έτσι ώστε να προστατευτούν τα ηχθίδια. Μετά η συνεργασία Νορβηγίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως έχουμε διαφορετικούς κανόνες, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα απορρίψουμε όλα επειδή υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες. Πρέπει να φροντίσουμε να κρατήσουμε αυτά στα οποία συμφωνούμε, να προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε ο ένα τον άλλον, ή εμεί την Νορβηγία. Μετά, όσον αφορά τι πρόσθετε ποσοστώσει, ισχύει ότι η εμει την ορβηγια μετα Επιτροπή έχει διαφορετική άποψη για τι ποσοστώσει, για τι επιπλέον ποσοστώσει. Και πώς αυτό συνδέεται με την απαγόρευση της απόρριψης αν θέλουμε βιώσιμη αλληλεία. δεν μπορούμε να αυξήσουμε την αλληλεία. Σωστά. Ο λόγος στην Κομισιόν για να διευκρινίσει τα πράγματα. Και μετά στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Καταρχάς, η ε, αυξήση των ΤΑΚ. Ο όρος ε, ΤΑΚ προκαλεί κάποια μικρή σύγχυση, γιατί επιτρέπει συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα, αλλά χρησιμοποιείται ουσιαστικά σήμερα για να σημάνει το συνολικό επιτρεπόμενη φόρτωση. Άρα μπορεί να φτάσει στο επιτρεπόμενο αλίευμα και να πετάξει το υπόλοιπο. Το θέμα είναι, που θέλουμε να εξασφαλίσουμε τώρα είναι ότι εκφορτώνεις ό,τι έχει κάνει σε ψαριά. Εάν το κάνει, τότε μπορεί να κρατήσει το ίδιο ποσοστό θνησιμότητα, αλλά με υψηλότερε εκφορτώσει. Αυτό που εννοούμε λοιπόν τώρα το ΤΑΚ είναι ότι πρόκειται να κρατήσει το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση δηλαδή μεταξύ των δύο ενιών του ΤΑΚ. Αυτό που θέλουμε είναι να εκφορτώνουμε οτιδήποτε αλλιεύεται. Αυτή τη στιγμή λέμε MSY στόχους σε επίπεδο TAC. Θέλουμε δηλαδή σίγουρα να θα σχηματίσουμε αυτό το οποίο απορρίπτεται, να το περάσουμε στο κομμάτι των εκφορτώσεων, χωρί όμω να αυξάνουμε τη θνησιμότητα των ηχθείων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ουσιαστικά έτσι ε, αναφέρεται πολύ ρητά στο σχέδιο σε ό,τι αφορά τους βακαλάους, γιατί λέει τις συνολικές ε, ε απομακρύνσεις από το αλίευμα μετά τις εκφορτώσεις και μετά ε, αφαιρούμε τις σχετικές απορρίψεις. Το πρόβλημα όμως είναι ότι έτσι δημιουργείται, μια ποσόστοση απόρριψης. Δηλαδή, ο αλλιέας αν έχει ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο και έχει εκφορτώσει τα πάντα, τότε συνεχίζει την απόρριψη. Οπότε στη, συνέχεια ε, είναι υψηλότερο το ποσοστό και έτσι δημιουργούμε ακόμη περισσότερε απορρίψει. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι εκφορτώνει οτιδήποτε αλλιεύει, αλλά δεν αυξάνει την θνησιμότητα πέρα από, το μέγιστο, από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα επιτρέπεται περισσότερα αλλιεύματα, περισσότερη, μεγαλύτερη ποσότητα εκφόρτωση, χωρί όμω να αυξάνεται η θνησιμότητα είναι ουσιαστικά για να μην δημιουργείται μία ε, σύγχυση μεταξύ αυτών δύο. Σε ό,τι αφορά τον χρόνο, συ, ε, δεσμευθήκαμε με Νορβηγία ότι θέλουμε να το πετύχουμε αυτό μέχρι το 2013. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε μόνο όταν είμαστε έτοιμοι. Ενδεχομένω να μπορούμε μόνο εν μέρη να το εξασφαλίσουμε αυτό και εν μέρη εννοώ τα τεχνικά μέτρα. Αναφέρθηκε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την επιλεξιμότητα για να μην αλλιεύονται πολύ μικροί νέαγνοι δηλαδή καταρχάς. Αλλά αυτό βέβαια και υπονοεί και μέτρα τα οποία θα μειώνουν ακριβώς και τα λίβματα στο Σκάγκερακ. Η Νορβηγία συμφώνησε πάνω σε αυτό. Εάν δεν καταφέρουμε να το εξολύσουμε το 2013 σε ό,τι αφορά την απαγόρευση απορρίψεων, τίποτα δεν σταματά τα κράτη-μέλη που ε, μπλέκονται σε αυτό να να λάβουν εθνικά μέτρα για να εισάγουν αυτά τα τεχνικά μέτρα, να βελτιώσουν την επιλεξιμότητα και να βελτιώσουν όλη κατάσταση ό,τι αφορά τις απορρίψεις εν αναμονή της, ε, του χρόνου που θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός. Και η Επιτροπή απογοητεύεται και το ότι κατά τα φαινόμενα θα έχουμε δυσκολία να πληρώσουμε τον ε, στόχο την ημερομηνία της 1ης πρώτου 2013. Το πρόβλημα μου είναι ότι ενδεχομένω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισάγουμε ε, μια απαγόρευση των απορρίψεων για του πέσουμε οι Πρέπει να βρούμε ε, νέα επίπεδα THC στη μέση του χρόνου και μετά να δουλέψουμε αναλογικά για το πότε θα πρέπει, πώς θα πρέπει να μειωθούν τα THC για το υπόλοιπο του εξαμήνου. Αυτό έχει λεχθεί και από το Κοινοβούλιο. Το ποιο θα πρέπει να είναι το όριο αυτό. Πρέπει πάντα να υπολογίζουμε πόσος χρόνος ε, απομένει για να εισάγουμε το μέτρο αυτό. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εισαχθεί στο μέσον του έτους. Αυτό που προσπαθούμε να αποφύγουμε λοιπόν είναι να υπάρχει μια καθυστέρηση με το 2014. Θα είναι απογοητευτικό αν πρέπει να περιμένουμε να καθυστερήσουμε το 2014. Αλλά βέβαια έχετε δίκιο ότι οι αλληλείς πρέπει να ξέρουν τι θα συμβεί το 2014. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η... το Δανέσκο Υπουργό Αλίας έχει ήδη ε, εισάγει ε, μέτρο και λέει ότι δεν θα υπάρχει απαγόρευση των απορρίψεων το 2014, αλλά θα συνεχίσουν ως έχει. Όμως η Επιτροπή ίσως μοναχικά, προσπαθεί να δει αν θα καταφέρει να εισάγει κάτι μέχρι το 2013. Δεν είναι ίσως ρεαλιστικό. Είναι μη ρεαλιστικό όμως να αρνηθούμε ότι φαίνεται εξαιρετικά πενιχρές οι πιθανότητε να γίνει, γιατί φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εν μέρει τα τεχνικά μέτρα μπορούν να εισαχθούν το 2013 ένα κομμάτι του που μπορεί να εισαχθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα ελέγχου, όπω είπα, η Επιτροπή απογοητεύτηκε ιδιαίτερα για το ότι η Νορβηγία δεν συμφωνούσε πάνω σε κοινά μέτρα ελέγχου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εισάγουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να εισάγουμε κάτι τέτοιο. σω να καταλήξουμε μια απαγόρευση απορρίψεων που θα ελέγχεται πολύ καλύτερα από ό,τι γίνεται από την Νορβηγία. Δεν θεωρώ όμω ότι αυτό είναι πρόβλημα. Η Νορβηγία επικρίνει επί χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την πολιτική περί των απορρίψεων. Καλό θα ήταν και εμεί να είμαστε επικριτικοί απέναντί του, εάν θεωρήσουμε ότι αυτοί από την πλευρά του δεν έχουν επαρκή μέτρα ελέγχου για την πολιτική περί απορρίψεων. Κατά εμά, η μη εισαγωγή σχετικών μέτρων από την Νορβηγία, που, μέτρων που είναι πολύ καλά για τον έλεγχο τη απόρριψη των ελευμάτων, δεν πρέπει να μα εμποδίσει εμά για να κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να εισάγουμε μια απαγόρευση μόνο στο χαρτί, στα χαρτιά και μετά να μην υπάρχει έλεγχο. Εάν θέλουμε να την εισάγουμε αυτό, πρέπει να γίνει σωστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Βόρεια Θάλασσα, ήμουν παρόν όταν συζητήθηκε αυτή η πρόταση. Βέβαια, αυτό ήταν όταν ήταν σχεδόν ολοκληρωμένη η, η... πρόταση και ενδεχομένως το ΡΑΚ ε, έχει μείνει περισσότερο στις φάσεις προετοιμασίας της πρότασης αυτής και θα ήθελε να συμμετέχει. Καθόλου τη διάρκεια του 2010 όμως ήταν μια σειρά ε, ομάδων εργασίας με την Νορβηγία που παρακολουθούσα και εγώ και που παρακολουθούσαν και, ε, παρακολουθούσε και η Νορβική βιομηχανία και η της Ευρωπαϊκής Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εξαιρετική εξαιρετικά επικοδομητική και χαίρεται πάρα πολύ για το ότι συμμετείχε η πλευρά τη Νορβηγία. συνεισέφερε τα μάλα στι τελικέ εκθέσει, πάνω στον οποίο βασίζεται ο κανονισμό αυτό. Ενδεχομένω ίσω να μην υπήρχε επίσημη διαβούλευση του ΡΑΚ στην περίοδο εκείνη, αλλά σίγουρα η βιομηχανία ε, ενεπλάκει πάρα πολύ ενεργά στι τεχνικέ συναντήσει, οι οποίε οδήγησαν συγκεκριμένη πρόταση. Και όπως είπα, και εγώ συμμετείχα σε συναντήσεις στο ΡΑΚ, όπου συζητήθηκε η πρόταση αυτή. Κάτι που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι υπήρξε κριτική ότι ίσως είμαστε υπερβολικά διαστικοί. Είμαστε διαστικοί όμως γιατί, και πιέζουμε γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε την συνέχεια της, ε, ε της συμμετοχής του Σκάγκεραγκ στην όλη συμφωνία. Η Νορβηγία ήθελε να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη τα οποία αλλιεύουν ε, στα χωρικά της ιδιωτέ θα πηγαίνουν και θα ακολουθούν τους νορβηγικούς κανόνες και όχι τους κανόνες του κράτους ε, σημαίας προέλευσης του αλλιευτικού σκάφους. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε την παραδοσιακή διασυνοριακή αλληλεία, και για το Σκάγκερακ. Θα πρέπει να έχουμε μια λύση και να έχουμε στο δυνατόν νωρίτερα κοινού κανόνε με την Νορβηγία. Ήδη εκπνέει όπου να είναι η ημερομηνία και γι' αυτό προσπαθούμε να εισάγουμε γρήγορα την πρόταση αυτή. Και αντί να περιμένουμε να εισαχούν τα πάντα με τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ, ίσω πρέπει να το δούμε αυτό σαν ευκαιρία. Να προσπαθήσουμε ε, να εισάγουμε τα μέτρα. Δεν είναι εύκολη άσκηση και υπάρχουν πάρα πολλοί άγνωστοι παράγοντε. Συνεπάγεται θεμελιώδη αλλαγή στην πολιτική μα και θα υπάρχει πάρα πολλή εμπειρία η οποία θα αποκομιστεί και λάθη τα οποία θα γίνουν και από τα οποία θα μάθουμε. Εάν πάντα όμως ε, ε, αναβάλουμε την οποιαδήποτε απαγόρευση, απορρίψεων μέχρι ότι λειτουργήσει τα πάντα τέλεια, τότε ποτέ θα λειτουργήσει τίποτα. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και η εμπειρία την οποία θα αποκομίσουμε από το Σκάγκερακ θα είναι πραγματικά πολύτιμη και για την ευρύτερη συζήτηση που θα γίνει σε ό,τι αφορά την απαγόρευση απορρίψεων σε άλλες περιοχές. Είμαι σίγουρος ότι οι λύσεις τις οποίες θα βρούμε σε κάθε περιοχή θα βασίζονται στην περιφερειακή συνεργασία με περιφερειακές ε, απαγορεύσεις που θα αντιμετωπίζουν ακριβώς τα περιφερειακά προβλήματα, τα προβλήματα συγκεκριμένων ζωνών. Αυτό το βλέπω λοιπόν σαν ευκαιρία για να ξεκινήσουμε. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα προς επίλυση, προσπαθούμε να το λύσουμε τον καλύτερα, δεν είναι τέλεια η κατάσταση, αλλά είναι πραγματική ευκαιρία για να αλλάξουμε τις ε, πρακτικές αλίες προς το καλύτερο. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίτμαν για διευκρινήσεις, όχι για περαιτέρω συζήτηση. Ε, και στο τέλος θα δώσω το λόγο στον κύριο Κούν για να κλείσουμε. Κύριο Βίτμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικές πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Έχει δίκιο η Κομισιόν. Ε, έγινε μια συνάντηση τεχνικής φύσεως, τεχνικής φύσεως, όπου συμμετείχαν οι ενδιαφερόμενοι της Αλίας, αλλά όχι κατά βάση εκπρόσωποι του ΡΑΚ. Συνεπώς δεν ήταν ευρείας εκπροσώπησης. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Οπότε, ε, ήμασταν παρόντες, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά στην πραγματικότητα δεν διαβουλεύτηκε κανείς μαζί μας επισήμως. Προφανώς, εμείς στο ΡΑΚ και στην ομάδα εργασίας έχουμε συζητήσει την κατάσταση στο Σκάιρα και το Κάτεγατ. Συζητήσαμε την πρόταση της Κομισιόν. Και σήμερα προσπάθησα να σας παρουσιάσω την άποψη των διαφορών μελών του ε, Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, αλλά το 1 τρίτο του ΡΑΚ αντιπροσωπεύει ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι οποίες δεν συμμετείχαν στις ε, συνεδριάσεις στις οποίες εξετάσαμε την πρόταση της Κομισιόν. Συνεπώς, κατά βάση, Εμεί εκπροσωπούμε μόνο ένα τμήμα του ΡΑΚ αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι που δεν ήταν παρούσε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ε, τώρα, για του τεχνικού κανόνε. Η, πρόταση, η Κομισιόν κάνει μια πρόταση ε, διμερή, να το πω έτσι. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη μεριά έχουμε την Ορβηγία. Πλην όμως, Ε, υπάρχει εντύπωση ότι θα περάσουμε από τα 90 στα 110 χιλιοστά ματιού. Η... Παρόλο που είναι θετικό, δεν οδηγεί σε βελτίωση της επιλεκτικότητας των δικτύων. Οι άλλοι θέλουν να συμμετάσχουν στην διαμόρφωση των κανόνων. Εμείς, ως ΡΑΚ, είμαστε πάντα στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης Κομισιόν αν θέλει να ακούσει τη γνώμη μας. Το ίδιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όταν οι, δουλειές, όταν οι εργασίες γίνονται εν αγνία μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κύριε Κούν, έχετε το λόγο να τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω εγκάρδια τον κύριο Βίτμαν από το Γνωμοδοτικό Συμβουλίο τη Βορεια Θάλασσα. Για μας είναι αποφασιστικής σημασίας να έχουμε τις πληροφορίες άμεσα για τα τεχνικά μέτρα και κατευθείαν από τους ε, εμπειρογνώμονες. Γι' αυτό λοιπόν συγχαρητήρια. Αυτό που θέλω να... αυτό που, στο οποίο θέλω να σκίσω κριτική όμως είναι στις καθυστερήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία σύνθηκη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Υπουργούς Αλίας και τρίτες χώρες ε, είναι σχεδόν έτοιμη να τεθεί σε ισχύ και την τελευταία στιγμή μας λέτε ότι πρέπει να το επιμηκύνουμε αυτό, ότι πρέπει να δώσουμε παράταση. Και είμαστε μονίμως υποπίεση. Και σε μια τέτοια περίπτωση όπου αποφασίζουμε για την κοινή αλληλευτική πολιτική για τα επόμενα 15 χρόνια ή 7. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Επίσης, και οι ψαράδες μας έχουν φτάσει στα ωριά τους όσον αφορά την ε, αλληλευτική πολιτική. Και σε λίγο κινδυνεύουμε να μην τα δεχτούν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι θα γίνει με, τις, ε, με τα αλλιεύματα, αν θα εκφορτώνονται, ε, τι θα γίνει με τις ποσοστώσεις, με την ανταλλαγή των ποσοστώσεων, με τις απορρίψεις, θα απαγορευτούν ή όχι. Όλε Κρίστενσεν τοποθετήθηκε ξεκάθαρα. Οι συνάδελφοι από το Γνωμοδοτικό Συμφούλιο τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα. Υπάρχουν, υπάρχουν οι προθεσμίες, υπάρχει η 1η Πρώτου 13, αλλά τι γίνεται. Οι συναδελφοι απο το γνωμοδοτικο συμφουλιο τοποθετηθηκαν ξεκαθαρα υπαρχουν υπαρχουν οι προθεσμιες υπαρχει η πρωτη η πρωτου 13 αλλα τι γινεται οι νορβηγοι μας λένε ότι θα το δεχτούμε μόνο αν αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν θέλουμε έλεγχο στα σκάφη και τώρα προσπαθούμε να ξεγλιστρήσουμε και να βρούμε κάποια λύση στη μέση και μας λένε καθυστερήσεις. Αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος. Χρειαζόμαστε βέβαια συζητήσεις, αλλά πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το πλαίσιο. Και οι ερωτήσεις που έθεσα και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι, δηλαδή τι θα γίνει εάν την 1η του 13 δεν έχουμε συμφωνία για τον κανονισμό ανάμεσα στην Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει, θα σταματήσουμε να ψαρεύουμε. Τι θα γίνει με τα τάκ, τι θα γίνει με, το, με τον μπακαλιάρο, με το γάδο. Δεν ξέρουμε. Δεν φτάνει να μας πιέζεται μόνο. Ένα πράγμα, και ένα πράγμα μπορώ να συστήσω. Εμείς ως ευρωβουλευτές να προσκαλέσουμε τα γνωμοδοτικά συμβούλια για να συνεργαστούμε έτσι ώστε να καταρτήσουμε μια σωστή αλληλευτική πολιτική. Τώρα όσον αφορά τον κανονισμό για τον έλεγχο πιστεύω πως από τη μία έχουμε είτε την απόρριψη είτε την συνολική εκφόρτωση. Τι χρειάζεται για να κάνεις μια σωστή αλληλεία. Ε, Χρειάζεσαι έλεγχο, χρειάζεσαι μέγεθος ματιού, χρειάζεσαι εκφόρτωση ή όχι εκφόρτωση και να ξέρεις τι γίνεται με τις απορρίψεις. Χρειαζόμαστε μέτρα ελέγχου για να καθορίζουμε τα μεγέθη. Πρέπει όλα αυτά να μπουν στον κανονισμό. Πρέπει να μπουν αυτές οι λεπτομέρειες. Διότι μόνο τότε μπορούμε να καταρτήσουμε μια αποδεκτή και σωστή αλληλευτική πολιτική. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ είπαν και ζήτησαν να μην πιεστούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να κάνουμε έναν σωστό κανονισμό. Μιλάμε για, για blue box, για ηλεκτρονικό έλεγχο, να υπάρχει εποπτεία στα αλληλευτικά σκάφη, στο πού αυτά αλλιεύουν. Μιλάμε για αυτόματη δορυφορική πλοήγηση. Ωραία. Κατανοητό. Μιλάμε δηλαδή για όλα αυτά και στεκόμαστε σε λεπτομέρειες. Στεκόμαστε, ξέρω εγώ, για τις κάμερες, ας πούμε, πάνω στα πλοία και το μέγεθος. Η κυρία Ρόντουστ μας είπε και πολύ σωστά είπε ότι αυτό θα αποτελέσει προηγούμενο για τον βασικό κανονισμό. Εάν δεν καταφέρουμε να κάνουμε έναν σωστό κανονισμό για το Σκάγερακ, θα καταποντιστεί και όλη η αληθική μας πολιτική και αυτό πρέπει να τα αποφύγουμε. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ όλους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τα μέλη του ΡΑΚ που ήταν μαζί μας σήμερα τους διερμηνείς. Ε, διακόπτουμε και συνεχίζουμε στις 3 το απόγευμα.